Chers collègues, je vous propose euh, euh, Μπορούμε να αρχίσουμε στο σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα να αναφέρω κάποιες τροποποιήσεις. Όσον αφορά τον απολογισμό της Σουηδικής Προεδρίας θα ακούσουμε σε λίγο τον κύριο Στίβ Ότο Λίτοριν, αλλά δεν θα τον συνοδεύει άλλη υπουργός γιατί την κυρία Χούσμαρκ Πέρσον δεν έχει τη δυνατότητα να είναι μαζί μας. Είναι υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων. Δεύτερη μεταβολή όσον αφορά την ανταλλαγή απόψεων όσον, για τη ρύθμιση όσων εκτελούν κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών θα δείτε ότι αυτό θα το κόψουμε σε δύο τμήματα. Αύριο το πρωί όταν θα αρχίσουμε τις εργασίες μας θα ήθελα και συμφωνήσαμε με την εισηγήτριά μας την κυρία Κούνστ ε, μία ενημερωτική παρέμβαση για το φάκελο των μικροεπενδύσεων να γίνει με την παρουσία των μελών της Επιτροπής. Αύριο το πρωί λοιπόν, ξεκινώντας τις εργασίες μας, η κυρία Κούνστ θα αναφερθεί σε αυτό το θέμα. Τέταρτη μεταβολή. Έχουμε την έκθεση πλόμπα. Τη βελτίωση της υγείας και της κοινωνικής ασφάλειας των εγγύων των λεχόνων και των γυναικών που θυλάζουν η συγγήτρια και διάφορα, διάφορες ομάδες μας ζήτησαν να μην ψηφίσουμε αύριο αυτή την έκθεση. Αναβάλλεται λοιπόν για την επόμενη συνεδρίαση για τις 27 Ιανουαρίου. Και αυτό μπορεί να γίνει εύκολα επειδή επί της ουσίας η Επιτροπή Γυναικών δεν θα αποφανθεί μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου. Τέλος μετά από αυτές τις τροποποιήσεις της μερίσιας διάταξης, σας παρακαλώ να μην αρχίσουμε αύριο το πρωί σε 9, αλλά σε 9.30. Ο κύριος Λέβιτσον. Είσαστε πολύ δραστήριο μέρος, μέλος, αναπληρωτής μεν, αλλά πολύ ενεργό μέλος. Σας δίνουμε λοιπόν αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να μεταφέρουμε τη συζήτηση για το σημείο 5 στον Ιανουάριο. Γιατί, κυρία Πρόεδρε, η συγκήτρια δεν είναι εδώ για το σημείο 5. Ελπίζω λοιπόν ότι μπορείτε να δεχτείτε να μεταφερθεί για τον Ιανουάριο η συζήτηση. Έτσι θα βελτιώσουμε το επίπεδο της συζήτησης με την παρουσία της συζήτητριας. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ναι, αυτό το αίτημα μου το διαβίβωσε η συγκήτρια και έχω μεγάλη συμπάθεια για την πολιτική της ομάδα. Όμως, αυτό το αίτημα μου υποβλήθηκε πολύ καθυστερημένα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι πολύ δύσκολο να, να κατασκευάσουμε την ατζέντα σημαίνει ότι θα πρέπει να διακόψουμε για τρία τέταρτα δεν μοιάζει λογικό αυτό αυτό το οποίο σας προτείνω και ελπίζω να υποστηρίξετε την πρότασή μου είναι το εξή. σήμερα να κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και όλοι θα σημειώ, πάρουν σημειώσεις για να αναφέρουν τις σχετικές παρατηρήσεις στην εισηγήτριά μας και πριν από την ψηφοφορία θα οργανώσουμε και δεύτερη ανταλλαγή απόψεων παρουσία της συγκύτρες έτσι θα έχει την ευκαιρία να διατυπώσει τις απόψεις της για τα διάφορα θέματα που θα έχουν τεθεί. Εν πάση περιπτώσει είναι πολύ κακή η πρακτική όταν έχουμε ένα τόσο σημαντικό φάκελο με τόσες τροπολογίες να ψηφίζουμε αμέσως μετά την παρουσίαση των τροπολογιών. Συνεπώς, Πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να έχουμε μια άτυπη ανταλλαγή απόψεων σήμερα για τις τροπολογίες και θα ξαναεντάξουμε στην ημερήσια διάταξη μελλοντικών συνεδριάσεων, θα βρει την κατάλληλη ημέρα η γραμματεία, για να έχουμε μια δεύτερη ανταλλαγή απόψεων, την παρουσία της εισηγήτριας, ώστε να οδηγηθούμε στους απαραίτητους συμβιβασμούς πριν από την τελική ψηφοφορία. Κύριε Λάτμιξον, ε, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Αλλά ζητά το λόγο, παρακαλώ. Να άκουσα το όνομά σας. Συμφωνώ σχετικά με την ιδέα σας να έχουμε μία αρχική συζήτηση σήμερα δηλαδή. Θα ήθελα όμως να υποβάλω και ένα άλλο αίτημα Αφήστε με να ολοκληρώσω με τον κύριο Λούντβινγκσον για να βεβαιωθώ ότι συμφωνεί με την πρότασή μου. Και μετά τα λέμε. Ο κύριος Λούντβινγκσον. Θα προτιμούσα πρέπει να σας πω να αναβάλουμε τη συζήτηση για τον Ιανουάριο. Είναι σημαντικό να συμμετέχει η συγγήτρια στη συζήτηση, αλλά τέλο πάντων, αν όλοι, όλα λειτουργήσουν σωστά και αποτελεσματικά, η πρότασή σας ε, εντάξει, μπορεί να έχει κάποια λογική. Αλλά παρόλα αυτά σας ζητώ, αν είναι δυνατόν, να αναβάλουμε. Η κυρία Κορνέλισον. Μια και δεν θα ψηφίσουμε αύριο το πρωί, μεταξύ 9 και 10, θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε αυτό το χρόνο για να προετοιμάσουμε τον τρίλογο και ε, αρχίσει η συνεδρίαση στις 10 και όχι στις 9. Να προετοιμάσουμε τον τρίλογο σας ζητώ για τις μικροεπενδύσεις, τις μικροχρηματοδοτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν χρησιμεύσε τίποτα ο Τρίλογος αύριο το πρωί, γιατί το Κορεπέρ συνεδριάζει αύριο. Από την τελευταία μας συνεδρίαση για τον Τρίλογο δεν έχουμε κανένα νέο στοιχείο, αναμένοντας τα αποτελέσματα του Κορεπέρ. Λοιπόν, ε, η ιδέα είναι να έχουμε μια συνάντηση, συνεδρίαση μάλλον, την επόμενη Δευτέρα Δευτέρα για να προετοιμάσουμε τον τρίλογο της επόμενης Τρίτης. Θα γίνει αυτό 8 με 9. 8 με 9 την Τρίτη, την επόμενη Τρίτη δηλαδή. Αύριο το πρωί λοιπόν θα ξεκινήσουμε τις εργασίες μας στις 9.30. Έχετε άλλα αιτήματα? Όχι. Προχωράμε λοιπόν και έχουμε πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό. Λυπάμαι που ο Υπουργό έπρεπε να παρακολουθήσει όλα μας τα πρακτικά, αλλά πώς να γίνει, χρειαζόμαστε να οργανωθούμε. Λοιπόν, ε, τα πρακτικά διανεμήθηκαν για 4 και 5 Νοεμβρίου, δεν υπάρχουν σχόλια, οπότε εγκρίνονται. Στο 3 τώρα έρχομαι, ανακοινώσει, αλλά θα τις αφήσω αυτές μετά την συνάντηση με τον Υπουργό. Συνεπώς, ευχαριστώ τον Υπουργό που είναι μαζί μας. Του δίνω αμέσω το λόγο. Το γεγονός ότι είστε σήμερα μαζί μας κάτω από δύο διαστάσεις θα έλεγα ε, δίνει ιδιαίτερο φως τη συμμετοχή σας. Πρώτα απ' όλα, σήμερα είναι η πρώτη μέρα της εφαρμογής της συνθήκης της Λισαβόνας. Ε, για μας, για τις υποθέσεις μας, έχει μεγάλη σημασία ιδιαίτερα το άρθρο 9 που μας δίνει αυτή την οριζόντια ρήτρα που σημαίνει ότι ό,τι σας ενδιαφέρουν και μας ενδιαφέρουν μπαίνουν σε άλλη ιεράρχηση όσον αφορά ε, την εφαρμογή ε, και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για δημόσιες υπηρεσίες ή ε, κοινού συμφέροντος. Θα έχουμε την ευκαιρία κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μας να επανέλθουμε σε αυτό και είναι πολύ σημαντικό όμως να υπογραμμίσουμε σήμερα ότι μπαίνουμε σε ένα νέο νομικό ορίζοντα και επίση πιστεύω ότι το γεγονός ότι ήρθατε να μας βρείτε σήμερα αφού συμφωνήσατε χθε για ένα φάκελο ο οποίο είχε μπλοκαριστεί και, ε, και αυτό είναι ένα πολύ καλό μήνυμα και σας δίνω τον λόγο για μια παρουσίαση που γνωρίζετε θαυμάσια πλέον γιατί έχετε συμμετάσχει ήδη όταν ήρθατε να μας δείτε στην αρχή της θητείας σας. Ο υπουργό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος όταν είναι ενδιαφέρον. Και πραγματικά είναι σαν να ήταν χθες που ήμουν πάλι κοντά σας το Σεπτέμβριο. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος τώρα της Σουηδικής Προεδρίας και χαίρομαι που είμαι εδώ για να ανασκοπήσουμε το έργο της Σουηδικής Προεδρίας στον τομέα σας και θα προσπαθήσω να αναφερθώ στα διάφορα θέματα ενδιαφέροντος. Λίγα λόγια εισαγωγικά όσον αφορά την αγορά απασχόλησης στην Ευρώπη σήμερα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η οικονομική και δημοσιονομική ε, κρίση έχει ε, σημαντικότατες επιπτώσεις στην απασχόληση. Η Ευρώπη θα χάσει πάνω από 7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας το 2009 και 10 και η ανεργία θα φτάσει το 10% το 2010. Αυτές είναι οι προοπτικές. Από τότε που ξεκίνησε η στρατηγική της Λισαβόνας έχουμε φτάσει στο 65,9% αλλά η σημερινή κρίση θα ανατρέψει αυτή την ανάπτυξη που έχει υπάρξει χάρη στη στρατηγική της Λισαβάνας. Αν και η κρίση είναι αισθητή παντού, οι επιπτώσεις είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Χθε είχαμε τη μοναδική συνάντηση ΕΠΣΚΟ κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας μαζί με την, ε, το, το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων. Και σήμερα, 1η Δεκεμβρίου, όπως είπε η Πρόεδρος, η συνθήκη της Λισαβόνας τίθεται σε, σε ισχύ και αλλάζει όλο το τοπίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί με όλες τις άλλες μεταβολές μέσα στην ΕΕ, πρέπει να λάβουμε μέτρα για να ανταποκριθούμε στις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση δεσμεύσεις, το μοίρασμα των εμπειριών μπορεί να μας οδηγήσει σε λύσεις ώστε η Ευρώπη να βγει διαρθρωτικά ισχυρότερη από την κρίση και καλά εξοπλισμένη για τις μελλοντικές προκλήσεις. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη συνάντηση έψκο χθε συζητώντας ακριβώς αυτά τα θέματα. Την τελευταία φορά που ήμουν μαζί σας το Σεπτέμβριο αισθάνθηκα ότι υπήρχε μεγάλη ανησυχία όσον αφορά την ευρύτερη κατάσταση και τους περιορισμούς που επιβάλλονται μέσω των μεθόδων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο για την απασχόληση. Άσχετα όμως με αυτό, πιστεύω ότι από διαφορετική προοπτική θα πρέπει να μην τα πάρουμε όλα τα θέματα σαν αριθμούς και ποσοστά, αλλά να σκεφτούμε τους ανθρώπους, τα άτομα, ε, με σάρκα και οστά που χάνουν τη δουλειά τους ή που δεν κατάφεραν ποτέ να μπουν στην αγορά εργασίας. Ε, είχαμε 100 εκατομμύρια Ευρωπαίους εκτός κανονικής αγοράς απασχόλησης πριν ξεκινήσει η κρίση. Ε, άνθρωποι που είχαν το, δίκαιο, το δικαίωμα μάλλον να ενταχθούν, να ζήσουν τα όνειρά τους, να λάβουν ένα μισθό, να, να είναι ενδιαφέροντες για τους άλλους και να επηρεάσουν και το μέλλον. Πριν από τρία χρόνια πήγα σε ένα πρόγραμμα στη Στοκχόλμη και συνάντησα έναν άνθρωπο που λεγόταν Λέι, δύο ετών νεότερος από μένα, με αναπηρική καρέκλα εδώ και 14 χρόνια, με σύνταξη και το μόνο που ήθελε είναι μια δουλειά, μια δουλειά να πάει να εργαστεί. Και πέραν όλων των στατιστικών και των αριθμών, περί αυτού πρόκειται. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται να γίνουν και αυτοί μέλη της κοινωνίας. Δεν είναι μόνο ζήτημα ανθρωπιστικό, είναι και οικονομικό ανάγκη. Δηλαδή, αν εξετάσουμε το μέλλον, έχουμε δημογραφικέ προκλήσεις σε όλη, την, σε όλη Ευρώπη. Αν θέλουμε λοιπόν να αναπτύξουμε το κοινωνικό μας σύστημα, να έχουμε σχολεία για το μέλλον, να έχουμε συντάξεις για τους περισσότερους από εμά μελλοντικά, πρέπει όλοι να συμβάλλουν. Ο κάθε Ευρωπαίος πρέπει να συμμετάσχει στην αγορά εργασίας για να επεκταθεί το κοινωνικό σύστημα. Μπορεί πολιτικά να διαφωνήσουμε πώς να οικοδομηθεί αυτό το σύστημα, πώς θα αναπτυχθεί κτλ. Αλλά δεν πρέπει να λείπει κανείς από αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό από την ώρα που τα εργαλεία στο επίπεδο της ΕΠΣΚΟ, το ευρωπαϊκό επίπεδο δηλαδή, ε, ο μηχανισμός αυτός περιορίζεται σε κάποια σημεία, γι' αυτό στο συντονιστικό ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να μπορέσουμε να παρέμβουμε σε οποιονδήποτε τομέα έχουμε αρμοδιότητα και να επιτύχουμε τη συμπερίληψη όλων. Θα έλεγα λοιπόν ότι η κοινωνική Ευρώπη ξεκινάει με μία δουλειά. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για συνοχή κοινωνική, η συμπερίληψη στην αγορά της εργασίας είναι ακριβώς αυτό. Ακόμη θέλουμε να εξασφαλίσουμε, να αποφύγουμε, να έχουμε μια αύξηση της ανεργίας που να οδηγήσει σε περαιτέρω αποξένωση. Ξέρουμε από τις προηγούμενες κρίσεις ότι όσα συστήματα και αν έχουμε είναι απαραίτητο να καταφέρουμε να μπει ο κάθε άνθρωπος πίσω στην αγορά εργασίας μόλις μπορέσουμε να επιτύχουμε τη μεταβολή πλήρης, το πλήρες δυναμικό εργασίας της Ευρώπης πρέπει να ενεργοποιηθεί για να εξασφαλίσουμε την επιμερία των πολιτών μας. Ε, ξεκινήσαμε βεβαίως με την άτυπη συνεδρία, συνάντησή μας στις αρχές Ιουλίου. Σας το είχα αναφέρει αυτό την προηγούμενη φορά που είχα έρθει. Ε, ένα από τα αποτελέσματα αυτής της άτυπης συνεδρίασης ήταν τα διάφορα ατομικά μέτρα που ελήφθησαν στα κράτη-μέλη ε, για να τεθούν σε ενέργεια, σε εφαρμογή τα καλύτερα εφικτά μέτρα για να αντιμετωπιστεί κρίση ώστε να οικοδομηθεί και μια υγιής μελλοντική Ευρώπη. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν αυτό το μικρό τετράδιο. Δεν θα σας εντυπωσιάσει σε μέγεθος, αλλά είναι η συλλογή των σωστών πολιτικών μέτρων από κάθε κράτος μέλος, ώστε να εξασφαλίσει να εξασφαλιστεί η παραμονή των, ε, στις θέσεις εργασίας ή η επιστροφή στην αγορά εργασίας το ταχύτερο δυνατόν. Υπάρχουν αντίγραφα αν σας ενδιαφέρει. Πολύ ωραία λοιπόν. Τα συμπεράσματα στον τομέα πολιτικής τα οποία καταλήξαμε χτες στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ ήταν τα εξή. Οι Υπουργοί Επασχόληση ε, άρχισαν να προετοιμάζονται για τα ζητήματα μετά τη Λισαβόνα. Τα συμπεράσματα πολιτική θα δοθούν στον Πρωθυπουργό μου και κατόπιν θα χρησιμοποιηθούν πριν την επερχόμενη Ισπανική Προεδρία για την διαμόρφωση της νέας ατζέντε μετά τη Λισαβόνα και θα επανέλθω στο σημείο αυτό κατόπιν. Είχαμε επίση ε, ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο που τόνισε ότι η πολιτική δέσμευση να ενεργοποιηθούν πολιτικέ ε, αγορά εργασία για να συνδέσουν την αγορά εργασία με την καινοτομία και να μειώσουν την ανεργία είναι κάτι αναγκαίο για να μπορέσει να υπάρχει μια μόνιμη χρηματοδότηση των δημοσίων οικονομικών Ξεκινώντας από τα συμπέρασμα του Συμβουλίου χτες, την πρόθεση της ένταξης στην αγορά εργασία, την αποκατάσταση, την ανάκαμψη από την κρίση και την προετοιμασία της ατζέντα του 2010 για το μετά τη Λισαβόνα. Το Συμβούλιο συζήτησε τα μέτρα που πρέπει να ρυθμούν σε κερδός οικονομική ύφεση για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τι αρνητικέ συνέπειε στην απασχόληση και το πώ θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται με τρόπο που θα μα επιτρέψουν να βγούμε από την κρίση διαφορετικά ισχυρότερη και καλύτερα εφοδιασμένοι για τους στόχους μας. Επίσης συζητήθηκαν τα στοιχεία της αγοράς εργασίας και τα στοιχεία κοινωνικής πολιτικής που οδηγούν στη δημιουργία καλύτερης, ε, πιο ε, πλήρων και ενσωματωμένων αγορών εργασίας. Το Συμβούλιο στη συζήτηση αυτή συμφώνησε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη συζήτηση. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα αυτά χρειάζεται να θεσπίσουμε ε, ισχυρότερη διαθωτικά αγορά εργασία για να εξασφαλίσουμε υψηλή απασχόληση, υγιή δημοσιοοικονομικά και μεγάλη ευημερία για όλου. Τα συμπεράσματα υπογραμμίζουν επίση ότι οι ενεργέ πολιτικέ αγορά εργασία και οι κοινωνικά δραστήριε πολιτικέ κοινωνική ασφάλιση είναι αναγκαίε για την ένταξη στην αγορά εργασία. Πιστεύω ότι τα συμπεράσματα αυτά δίνουν σαφέ μήνυμα προ το δεκεμβριανό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την επερχόμενη Ισπανική Προεδρία και θα συμβάλλουν συζητήσει για τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τι θέσει εργασία και τη δουλειά μετά το 2010. Να σα τονίσω επίση ότι αναγνωρίζω πω ε, η Προεδρία μα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ε, Είχαμε ένα εκλεγέν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είδαμε μια ανανέωση των συνθήκων, κάτι που ολοκληρώθηκε φέτος είχαμε μία απελθούσα επιτροπή. Περιμένουμε ακόμα το να ξεκινήσουν οι νέοι επίτροποι. Δηλαδή, κάναμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε για να πετύχουμε αυτή την Προεδρία, αφήνοντα στην Ισπανική Προεδρία αρκετή δουλειά ακόμα. Και στην Κομισιόν. Περιμένω λοιπόν τώρα και καλό συντονισμό και στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα που μας απασχολούν. Σας χρειαζόμαστε, χρειάζεται ο ένας τον άλλον για να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε ένα σωστό μέλλον μπροστά μας. Όπως είπα πριν από λίγο, τον αντίκτυπο της κρίσης τον αντιμετωπίζουν τον υφίσταται κυρίως άνθρωποι. Και μία πρόταση μείωση του αρνητικού αντικτύπου είναι η πρόταση της για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δομή διευκόλυνση μικροχρηματοδότηση. Μια βελτίωση της ε, ευκολία πρόσβασης στη μικροπίστη μπορεί να ενισχύσει την δημιουργία μιας ε, αγορά εργασία με μεγαλύτερη συμμετοχή όλων. Όλοι θεωρούμε ότι πρέπει να βελτιωθούν οι εργασιακές προοπτικές των πληγέντων από την κρίση. Και τα βασικά στοιχεία τη πρόταση αυτή ήταν προτεραιότητα για μα. Ελπίζω να συνεχιστούν. Όπω ξέρετε, συζητούμε με το Κοινοβούλιο το δοσιέ κατά τη κρίση. Όπως ξέρετε, το προσεπίληση ζήτημα αφορά τη δημοσιονομική διάσταση της πρότασης και τη χρηματοδότηση του μέσου αυτού. Το Συμβούλιο υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να φύγουν κονδύλια στο νέο, στη νέα διευκόλυνση από το εφιστάμενο πρόγραμμα χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και ελπίζουμε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη, το κείμενο σε πρώτη ανάγνωση. Α το ευχηθούμε. Γιατί πρέπει να σας πω ότι δεν είναι εύκολο ζήτημα. Πιστεύω ότι η επίτευξη συμφωνία στο εργαλείο αυτό, για το εργαλείο αυτό δεν είναι ένα πρώτο σαφέ βήμα μια Ευρωπαϊκή συγκεκριμένη πολιτική καταπολέμησης τη κρίση. Ελπίζω να περάσει αυτό μέσα στην Προεδρία μας. Έχουμε ακόμα ένα μήνα. Άλλο ζήτημα. Ο συνδυασμός οικογενειακής και εργασιακής ζωής. Χτες το Συμβούλιο δέχθηκε μια ε, νέα οδηγία για τη γονική άδεια που ενισχύει τη δυνατότητα των γονέων, μητέρων και πατέρων να συνδυάζουν την εργασιακή τους ζωή με την οικογενειακή ζωή. Επίσης, ε, η Επιτροπή Γυναικών ε, του Κοινοβουλίου υποστηρίζει την συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους και το σχέδιο ψηφίσματος για την εξισορρόπηση του οικογενειακού, της οικογενειακής ζωής και της ε, εργασιακής ζωής. Η πρόθεση της ισότητας των φύλων επιτρέπει και η βοήθεια στις γυναίκες για να συνδυάσουν οικογενειακή και επαγγελματική ζωή είναι προτεραιότητα για μας, γι' αυτό πετύχαμε πολιτική συμφωνία για την οδηγία για τις αυτοπασχολούμενους χτες στο Συμβούλιο έψκο. Η Προεδρία είχε επίση την πρόθεση να συνεχίσει να δουλεύει στην οδηγία για την μητρική άδεια και να προχωρήσει τι διαπραγματεύσει σχετικά ε, στην άδεια μητρότητα, συγγνώμη, και να προχωρήσει τι οδηγίε στο ταχύτερο δυνατό. Ε, συνεργαζόμαστε με την εισηγήτρια του Κοινοβουλίου, κυρία Στρέλα, για το χρονοδιάγραμμα για το Κοινοβούλιο. Ο Υφυπουργό Απασχόληση τη Σουηδία μετέσχε σε μια συζήτηση για την οδηγία και για την συζήτηση για την διαλογή οικογενειακής και επαγγελματική ζωή που έγινε στην Επιτροπή στι 4 Νοεμβρίου. Επιπλέον, ο Υπουργό Ένταξη και Ισότητα Φίλων τη Σουηδία επισκέφθηκε το φθινόπωρο την Επιτροπή Γυναικών. Περιμένουμε τη νέα έκθεση τη Επιτροπή και οι συνεργασίε για την πρόταση αυτή συνεχιστούν και επί Ισπανική Προεδρία. Η διάσκεψη υψηλού επίπεδου για την ένταξη στην αγορά εργασία 26-28 Οκτωβρίου ήταν επίση μια καλή ευκαιρία για να συγκεντρωθούν πολιτικοί, ειδικοί και άλλοι εμπλεκόμενοι φορεί για να συζητήσουν πολιτικέ για την καταπολέμηση τη κρίση των θέσεων εργασία, χωρί να τεθεί σε κίνδυνο ο μακροπρόθεσμο στόχο και η δημιουργία μια ισχυρή Ευρώπη στο μέλλον. Η διάσκεψη προσέφερε παρουσίαση νέων ενδιαφερουσών μελετών και συζητήσει για διάφορε πτυχέ ε, ένταξη στην αγορά εργασία. Μία από τι συνόδου ασχολήθηκε με τον εντοπισμό των δράσεων που χρειάζονται για να υπάρξει συμμετοχή, ε, ποσοστό συμμετοχή ε, του εργατικού δυναμικού που θα εξασφαλίζει την ευημερία όλων των πολιτών τη Ευρώπη. Μια άλλη σύνοδο ασχολήθηκε με τι βασικέ προκλήσει που αντιμετωπίζει η αγορά εργασία τη Ευρώπη την επόμενη δεκαετία, ενώ η τρίτη σύνοδο ασχολήθηκε με το πώ μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση στην απασχόληση μέσω ενεργικού ε, κοινωνική πολιτική και πολιτική κοινωνική ασφάλιση. Παράλληλα με την σύνοδο, έγινε και ένα υπουργικό εργαστήρι για να δώσει στους υπουργούς την ευκαιρία να συζητήσουν πόσο θα διαχειριστούν τον αντίκτυπο των, της οικονομικής και κλιματοοικονομικής κρίσης με, αυξάνοντας την πρόσβαση στην απασχόληση. Οι συζητήσεις ε, περιστράφηκαν γύρω από εθνικά μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση των, της κρίσης και έγινε ανταλλαγή καλών εμπειριών of the Swedish presidency. And I'm sure that... Έχει ακόμα ένα μήνα η Σουηδική Προεδρία. Ελπίζω να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις υπόλοιπες προκλήσεις πριν στο τέλος του μήνα δώσουμε την Προεδρία στην Ισπανία. Θέλω σε προσωπικό επίπεδο να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Απασχόληση για την συνεργασία σας στους τελευταίους μήνες. Περιμένουμε να συνεργαστούμε μαζί σας και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Κάνατε μια καλή παρουσίαση για μια προεδρία που ζούσε σε δύσκολο χρονοδιάγραμμα μεταξύ δύο κολεγίων επιτρόπων, μιας ε, προσεπικ... διαδικασία ε, διαδικασίας και με αποτελέσματα αρκετά θετικά χάρη στις θέσεις στο Συμβούλιο. Υπάρχουν βεβαίως και άλλα εκκρεμή ακόμα ζητήματα, κρίσιμα μερικές φορές μεταξύ των δύο οργάνων. Πιστεύω ότι είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουμε στις συζητήσεις που έχουμε τώρα. Δίνω το λόγο στην κυρία Κίνγκερ Κούντς, η συγγήτριά μας όπως όλοι γνωρίζετε, για το σχέδιο για την μικροπίστωση. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τα σχόλιά σας και για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την επιτυχία σας. Ξέρουμε ότι ήταν δύσκολη η μήνες της Προεδρίας σας, ε, εν το μέσο κρίσης. Είναι δύσκολο να είναι κανείς υπουργό ε, Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης. Συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα είπατε. Είπατε ότι όντω, ε, παρόλο που βλέπουμε κάποια σημάδια έτσι ανάκαμψης ε, στην Ευρώπη αυτό που προβλέπετε είναι να χειροτερεύσει η κατάσταση της απασχόλησης. Νομίζω αναφέρατε ότι περιμένουμε ακόμη 2 εκατομμύρια άτομα ανέργων το 2010 και ένα ρυθμό ανεργίας αυξανόμενο μέχρι το 10% που είναι ούτως ή άλλως πολύ ψηλό σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης αναφέρατε ότι μιλούμε για ανθρώπινη ζωή, δεν είναι στατιστικά οι άνθρωποι αυτοί, είναι άνθρωποι. Και χρειαζόμαστε τους πάντες έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει ανάκαμψη στην Ευρώπη στα επόμενα χρόνια. Σημαντικό είναι ότι η κοινωνική Ευρώπη ξεκινά με την απασχόληση. Και αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω ή να σας ζητήσω την δέσμευσή σας, την υποστήριξή σας για αυτά τη δυνατότητα μικροχρηματοδότησης που μπορεί όντως να είναι ε, μεγάλη επιτυχία για την ε, ε, Σουηδική Προεδρία και υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε σε μία λύση αν και μερικέ φορέ δεν κατάλαβα ακριβώ γιατί αυτέ οι, δια... οι διαπραγματεύσει ήταν τόσο δύσκολε, γιατί από όσο κατάλαβα εγώ, όλοι συμφωνούσαν ότι αυτό είναι κάτι που χρειαζόμαστε. Όλοι ξέρουμε ότι όσοι χάνουν τι ε, θέσει εργασία του, χάνουν και τι ικανότητέ του και δεν είναι τόσο εύκολο να επανέλθουν μετά από κάποιου μήνε, έξι μήνε, ένα χρόνο στην αγορά εργασία. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε ένα είδος, ένα μέτρο, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να παραμείνουν ενεργοί για να επιστρέψουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην αγορά εργασίας. Να τους βοηθήσουμε όχι μόνο οικονομικά, αλλά με συμβουλές, με υποστήριξη για να μάθουν να, να ενισχύσουμε τις ικανότητές τους. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσει η Σουηδική Προεδρία ε, να πιέσει για το πρόγραμμα αυτό, γιατί εμείς θεωρούμε ότι ήταν πραγματικά πολύ επιτυχές. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο. Γι' αυτό ελπίζουμε να μπορέσετε να πιέσετε και το Συμβούλιο. Να... Το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να υποστηρίξει το πρόγραμμα αυτό όσο μπορούμε να το κάνουμε. Πραγματικά χρειαζόμαστε όμως και την υποστήριξη του Συμβουλίου και της Σουηδικής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα. Είμαστε ε, και οι δύο και στο ίδιο, στην ίδια πλευρά είμαστε και οι δύο. Κατανοούμε ότι αν θέλουμε να υπάρξει συμφωνία, φυσικά πρέπει να υπάρξει και κάποιο συμβιβασμό. Ε, έτσι γίνονται τα πράγματα συνήθω. Το πρόβλημα που βλέπουμε είναι ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα δημοσιονομικά και εκεί έγκυται το πρόβλημα. Πιέζουμε ε, για να, βρεθεί μια ισορροπία και αν μπορώ και εγώ να σας ζητήσω ε, να μιλήσετε με τα Υπουργεία Οικονομικών σας και να ε, τους πείτε να χαλαρώσουν λίγο γιατί θα μας βοηθούσε πολύ. Φυσικά θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό το συντομότερο δυνατό γιατί όταν θα καταφέρουμε ε, να επιτύχουμε την, την συμφωνία μπορεί η κρίση να έχει τελειώσει αν να καθυστερήσουμε κι άλλο. Φοβούμαι ότι στη φάση αυτή υπάρχει περίπτωση να υπάρξει μια μικρή μειοψηφία στο Συμβούλιο που θα μπλοκάρει την όλη προσπάθεια. Ελπίζουμε να μην γίνει αυτό. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Θα είμαστε σε επαφή. Εγώ συνεχώς προσπαθώ να πείσω τους συναδέλφους μου έτσι ώστε και αυτοί να πείσουν τους δικούς τους συναδέλφους στην κυβέρνηση να δεχτούν. Αλλά όντως χρειάζεται στενή συνεργασία και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Να είστε βέβαιος ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα... Είμαστε βέβαιοι ότι θα χρησιμοποιήσετε όλα αυτά τα επιχειρήματα και στους υπόλοιπους υπουργούς μέχρι μεθαύριο προσπαθώντας να πείσουν τους άλλους υπουργού. Η πρόταση που κάνετε είναι λογική και νομίζω ότι όλοι θέλουν στην Επιτροπή να πετύχει η διευκόλυνση για τις μικροπιστώσεις και γρήγορα μάλιστα υπό τη δική σας προεδρία. Πρέπει να πείστε λοιπόν όχι μόνο τους Υπουργούς Κοινωνικών Υποθέσεων αλλά και τους Υπουργούς Οικονομίας. Η κυρία Μωρά και μετά η κυρία Μίλη Τούρινεν. Κύριε Μωρά, ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό που ήρθε ακόμα μία φορά για να μας ενημερώσει για την πορεία των εργασιών κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας. Δεν θα προσθέσω τίποτα σε αυτά που αναφέρθηκαν για την ε, μικροπίστωση. Ξέρετε ότι όλοι συμφωνούμε με την άποψη αυτή. Η προσωπική πρωτοβουλία είναι η πηγή της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Όσο μικρό, μικρή λοιπόν να είναι η χρηματοδότηση, πάντα είναι μια σημαντική συνεισφορά να συμβάλλουμε στην δημιουργία θέσεων εργασίας. Θέλω να σταθώ σε δύο σημεία που θεωρώ σημαντικά στην προσπάθειά μας να καταπολεμήσουμε και τις συνέπειες της κρίσης αλλά και τα προβλήματα απασχόλησης εν γέννη. Με δύο ερωτήματα που αφορούν την ενεργή ένταξη μέσω της απασχόλησης. Πώς βλέπετε το ενδεχόμενο να μπορέσουμε υπό τη δική σα Προεδρία να επιταχύνουμε την ένταξη των νέων στην αγορά εργασία. Ξέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της κρίση, οι νέοι που τελειώνουν τι σπουδέ τους είναι αυτοί που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία, από την κρίση και που αντιμετωπίζουν σοβαρές, σοβαρότερες δυσκολίες. Μπορούμε βέβαια να θέτουμε μεγάλους στόχους μάχης κατά της ανεργίας, αλλά οι νέοι είναι ένας πληθυσμός ιδιαίτερα ευάλωτος. Τι κάνουμε με τους νέους αυτούς που παλεύουν μάτια να μπουν στην αγορά εργασία. Μέσα σε αυτούς τους νέους δε υπάρχει μια ακόμα πιο ευάλωτη ομάδα. Οι άνθρωποι που μπαίνουν στην αγορά εργασία χωρίς προσόντα η έλλειψη επαγγελματικών προσόντων είναι ένας μόνιμος παράγων κοινωνικής αποσταθεροποίησης. Έχετε κάποιο στόχο ειδικό για αυτούς τους νέους, χωρίς προσόντα. Ένα ακόμα θέμα. Μιλήστε για ένα δίκτυο ασφαλείας για να επανέλθει κανείς στην αγορά εργασίας δημιουργήσαμε όλοι ένα εξαιρετικό εργαλείο, την επικύρωση των, και, των, της εμπειρίας. Αλλά ξέρουμε ότι το εργαλείο, το κουτί αυτό με τα εργαλεία δεν προχωράει γρήγορα. Σκέφτεστε την, το ενδεχόμενο επιτάχυνσης της διαδικασίας επικύρωσης των δεδομένων των, των, της εμπειρίας, της, της ε, εμπειρίας. Ευχαριστώ. Η κυρία Τούρινεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Υπουργό που έρχεται για δεύτερη φορά. Όντως δίνουμε έτσι το σωστό μήνυμα. Έχω ένα ερώτημα. Όταν μιλούμε για το καθεστώς, κοινωνικό καθεστώς και καθεστώς απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε λίγο την συζήτηση, να δείξουμε αισιοδοξία, όχι απεσιοδοξία. Και πραγματικά το λέω αυτό γιατί όταν ε, ακούω ε, επιχειρηματίες, ε, συνδικαλιστές, μου λένε ότι είναι άσχημη η κατάσταση και είναι πραγματικά πολύ δύσκολο τα πράγματα. Είναι, ε, υπάρχει το θέμα των, ε, το, της μισθοδοσίας, υπάρχει το θέμα των, ε, των θέσεων εργασίας στο εξωτερικό, υπάρχει ούτως ή άλλως και πολύ κοινωνικό ντάμπινγκ και πρέπει να υπάρξουν θαραλέοι πολιτικοί οι οποίοι όντως θα χτυπήσουν το πρόβλημα στη ρίζα του. Τα συνδικάτα είναι πολύ θετικά έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δανία και για μας είναι δύσκολο να τους εξηγήσουμε γιατί δεν βελτιώνεται η κατάσταση. Θα ήθελα να μου πείτε τι έκανε πραγματικά η Σουηδική Προεδρία ως προς αυτό, για το κοινωνικό ντάμπινγκ δηλαδή και για την απόσπαση εργαζομένων σε άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Thank you very much. Εγώ ευχαριστώ. Να ξεκινήσω απαντώντας στην κυρία Μωρά ε, για την αγορά εργασίας. Όντω υπάρχει μεγάλη αναστάτωση σε ό,τι αφορά το γεγονό ότι πολλοί νέοι έχουν πολλά προβλήματα να μπουν στην αγορά εργασία. Αν δείτε με το πέρασμα του χρόνου και ανεξάρτητα από την χώρα και ανεξάρτητα από τα συστήματα, ε, τα οργανωτικά και τα συστήματα κοινωνικής, ε, ε, τα κοινωνικά συστήματα, θα δει κανείς ότι οι νέοι σε όλες τις χώρες τείνουν να επιδεικνύουν ε, ε, διαφορετικές τάσει. Όταν ε, δηλαδή η κατάσταση χειροτερεύει είναι οι πρώτοι που φεύγουν από την αγορά εργασία, Όταν τα πράγματα ανακάμπτουν είναι οι πρώτοι που έχουν την δυνατότητα να έχουν θέση εργασία. Η κατάσταση τώρα στη ΣΥΠΑ α πούμε είναι περίπου στο 9% η, η ανεργία και η ανεργία των νέων είναι περίπου διπλάσια. Πραγματικά λοιπόν είναι πολύ διαφορετικές οι καταστάσεις ε, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και στην ε, Ευρώπη και σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και σε ό,τι αφορά την αγορά εργασία. Θεωρώ όμω ότι αν δούμε τις χώρες που ήταν πιο επιτυχεί στο να κρατήσουν ε, σε κάποια όρια την ανεργία των νέων, Δύο λέξεις θα μπορούσαν να περιγράψουν την κατάσταση αυτή. Ενεργοποίηση και εκπαίδευση ενεργοποίηση, δηλαδή να προσπαθήσουν να διατηρήσουν, να κρατήσουν τους νέους όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αγορά εργασίας ακόμη και όταν υπάρχει ύφεση. Και εκπαίδευση, όπως είπατε και εσείς κυρία Μωρά, είναι πάρα πολύ σημαντικός τομέας για να προετοιμαστούν οι νέοι για να μπουν στην ε, αγορά εργασίας, να ενταχθούν στο εργασιακό τους περιβάλλον. Και πέρα από αυτό, οι χώρες θεωρώ ότι ε, λίγο πολύ τα καταφέρνουν στο να έχουν στενή σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων και της αγοράς εργασίας. Αν ας πούμε πάμε στη Δανία ή στις κατοχώρες. Νομίζω ότι θα δείτε πως ε, έχουν αρχίσει οι σχέσεις να γίνονται πιο στενές και οι επαφές πιο πολλές μεταξύ των ακαδημαϊκών ε, συστημάτων και της αγοράς εργασίας. Ας πούμε, εμείς δεν έχουμε τόσο καλές σχέσεις στην Σουηδία. Και αυτό πραγματικά είναι μειονέκτημα δικό μας, γιατί πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι, πολλοί νέοι φεύγουν, ε, τελειώνουν το σχολείο, χωρίς όμως να έχουν καμία επαφή με την αγορά εργασίας. Και ο Όλε Λούντβιξον ε, ήταν ε, στην Σουηδία πολύ ενεργό συνδικαλιστή και το δικό του, του, το δικό του συνδικατό πραγματικά είχε πολύ καλέ σχέσει στο να προσπαθήσει να ενισχύσει την αγορά εργασία, να μπουν οι νέοι πιο οργανωμένα στην απασχόληση. Και Υπάρχουν πολλά τέτοια καλά παραδείγματα. Μπορεί αυτό να γίνει μέσω της, ε, των εκπαιδευτικών συστημάτων, μέσω των κοινωνικών εταίρων έτσι ώστε να υπάρξουν αυτοί οι δεσμοί μεταξύ των ακαδημαϊκών και των επιχειρηματιών. Αυτό είναι ένα από τα σημεία κλειδιά που πρέπει να προσέξουμε. Τώρα, σε κάποιες άλλες χώρες θα σας πούνε κάτι διαφορετικό. Στη Δανία ίσως σας πούνε ότι υπάρχουν και οικονομικά θέματα. Βέβαια, εντάξει, αυτό δεν θέλω να το θίξω τώρα, αλλά... Αν δούμε το κοινωνικό dumping, διστάζω, δεν μου αρέσει αυτό αυτός ο όρος. Καταρχήν, γιατί δίνει ένα μήνυμα ότι το να μετακινηθεί κανείς από τη μια χώρα στην άλλη είναι κακό, είναι άσχημο. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Γενικώ είναι καλό το να έχει κανείς τη δυνατότητα να αποσπάται από τη μια χώρα στην άλλη και να εργάζεται εκεί. Είναι καλό. Ε, ως Σουηδός, αν μπορώ να μιλήσω, αυτό θα σας πω. Αν δούμε τα δημογραφικά στοιχεία, ε, χρειαζόμαστε πάρα πολλούς αν δούμε ας πούμε τι θα γίνει σε 10, 20, 30 χρόνια. Οπότε νομίζω ότι γενικώ οι αποσπάσεις είναι καλές και κερδίζει κανείς νέες εμπειρίες. και για τον ίδιο αλλά και για την αγορά εργασίας. Παρ' όλα αυτά, όπως θα θυμάστε, όταν, όταν ε, υπήρξε η απόφαση του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πραγματικά ήταν ατυχής και αυτό ήταν το πρώτο ε, σχόλιο που είχα κάνει για μια σχετική υπόθεση. Η δική μας θέση, η αρχική, ήταν ότι στη Σουηδία θα πρέπει να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις σουηδικές και σχετικοί κανονισμοί ω προ αυτό. Αλλά τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την νέα κατάσταση, πρέπει να τη διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο, όπω ο καλύτερο μπορούμε. Είχαμε την ε, ε, έρευνα Λαβάλ που ε, προέκυψε, από την οποία προέκυψε μία πρόταση, την οποία υποβάλαμε στο Κοινοβούλιο, παρουσιάστηκε πριν από λίγους μήνες. Ήταν η καλύτερη ισορροπία που μπορούσαμε πούμε, να βρούμε. ώστε να μην χρειάζεται με τον νόμο να επιβάλλουμε ελάχιστους μισθούς στην Σουηδία. Και υπάρχει ακόμα κάποια, κάποιο περιθώριο για τις συλλογικές συμβάσεις με κάποιες προϋποθέσεις που σχετίζονται και με την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Είναι όντως πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό για όλους και πιστεύω ότι η Κομισιόν έχει κάνει καλή δουλειά προσπαθώντας να βελτιώσει τη διαφάνεια. Όντω συνεργάζονται πολύ στενά και με του κοινωνικού εταίρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί την τελευταία φορά. Δύο στοιχεία έχουν υπάρξει στην συζήτηση για τις κοινωνικές ρήτρε που σχετίζονται με την συνθήκη. Εντάξει, τώρα είναι αργά βέβαια γι' αυτό. Από σήμερα ξεκινά να ισχύει η Λισαβόνα, οπότε αυτό το τρένο το χάσαμε. Το δεύτερο στοιχείο είναι να γίνει μια αναθεώρηση της οδηγίας για τις αποσπάσεις. Ξέρω ότι ο πρόεδρος Μπαρόσο έχει μιλήσει για ένα είδος ε, εφαρμοστικού κανονισμού. Δεν είμαστε ακριβώς σίγουροι τι θα πει αυτό. Δεν ξέρω εσείς κυρία Πρόεδρε αν ξέρετε. Αλλά πραγματικά περιμένουμε την Κομισιόν να μας απαντήσει ως προς αυτό για να δούμε τι ακριβώς είναι. Η αλλαγή τώρα για τις οδηγίες για τις αποσπάσεις, η αναθεώρησή της. Το συζητήσαμε την προηγούμενη φορά. Ας δούμε καταρχήν τι θα μας πει η Κομισιόν. Ε, είναι αρκετά ευαίσθητο το θέμα ε, και είναι και σημαντικό να ξέρει κανείς τι λένε οι κανονισμοί, να ξέρουν από πριν τι, πρέ, τι μπορεί να περιμένει και να μπορούμε μετά να δράσουμε αναλόγως και αποφεύγω το κοινωνικό ντάμπινγκ, αποφεύγω αυτούς τους όρους γιατί όντως δεν θέλουμε φυσικά να υπάρχει διακριτική μεταχείριση στην, ε, στην αγορά εργασία μετά από την απόφαση του δικαστηρίου. Πρέπει να υπάρχει μια τάξη στο σύστημά μας. Αν απαντώ έτσι στο ερώτημά σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοφεράτη και μετά η κυρία Πασκάλ Γκρονή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, όπως είπατε, και όπως έκανε και η Προεδρία σας αυτούς τους μήνες, να δουλέψετε για την αύξηση της αγοράς εργασίας σε μια κατάσταση βαθιάς κρίσης, όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Οπότε οι ρυθμίσεις για τη γονική άδεια, η βοήθεια στις μητέρες που θέλουν να κάνουν ένα παιδί, όλα όσα δημιουργούν ισοτήρια τη μία μεταξύ των φύλων βοηθά και στην αύξηση της αγοράς της εργασίας. Η αγορά εργασίας ωστόσο επηρεάστηκε και ποιοτικά, διότι η έκθεση πολλών, η, η απομάκρυνση πολλών ατόμων από την αγορά εργασία, ιδιαίτερα με την πρόοδη συνταξιοδότηση, οδηγήσε σε μια συνολική απώλεια γνώσεων. Οι γνώσει και ο επαγγελματισμό δεν συνδέονται πάντα με την πορεία και την ηλικία των ατόμων. Είναι όμως προφανές ότι όσο περισσότερο προχωρούν στη δουλειά τους οι άνθρωποι, τόσο μεγαλύτερη εμπειρία, αν όχι επαγγελματισμό, αποκτούν. Δεν πιστεύετε λοιπόν ότι είναι σημαντικό να συνοδεύσουμε τις ρυθμίσεις για την αγορά εργασία με παράλληλες ρυθμίσεις για την κατάρτιση, με ειδικά προγράμματα που θα στοχεύουν στην επανικοδόμηση του επαγγελματισμού που χάθηκε. Για το ντάμπινγκ τώρα. Πιστεύω όπως και εσείς ότι οι διαδικασίες κινητικότητας των νέων ιδίως πρέπει να θεωρηθούν θετικές. Μην ξεχνάτε όμως την διαφορά μεταξύ ενός νέου που μπορεί να επιλέξει που να πάει και σε μια χώρα μακριά από τη δική του και ενός ανθρώπου που είναι υποχρεωμένος να μεταναστεύσει γιατί δεν έχει εναλλακτική λύση. Στην περίπτωση αυτή δεν πιστεύετε ότι για το μέλλον, ιδίω μετά την έξοδο από την κρίση, είναι σημαντικό ταυτόχρονα με τη διαχείριση της αγοράς εργασίας να υπάρχει και ένα συντονισμός των αναδιανεμητικών πολιτικών, διότι για, τον ίδιο, ε, για τα ίδια επαγγέλματα και η δυναμική του κόστου της προσφοράς μπορούν να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις σημαντικές στο εσωτερικό της ίδιας χώρας και μεταξύ χωρών. Τώρα, μια διαχείριση αποκλειστική της αγοράς εργασίας, ανεξάρτητα από τον συντονισμό των φορολογικών πολιτικών και των μισθολογικών γενικότερα, μπορεί να είναι χρήσιμο, αλλά όχι επαρκές. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρονή. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, Μπορείτε να μα διαβεβαιώσετε ότι το θέμα τη απασχόληση θα είναι προτεραιότητα στην επόμενη Σύνοδο Κορυφή του Δεκεμβρίου. Από ό,τι είπατε, είναι ένα θέμα που και εσεί και εμεί θεωρούμε πολύ σημαντικό για την κρίση. Στα συγκεκριμένα μέτρα που προτείνεται, συμφωνώ και αυτά που είπε ο συνάδελφο για του νέου, αλλά εγώ έχω ένα άλλο θέμα που με ενδιαφέρει. ή Τα άτομα με αναπηρίες που αποκλείονται ακόμα περισσότερο. Έχετε συγκεκριμένα μέτρα. Μετά, οδηγία για την υγιεινή και ασφάλεια των γυναικών ε, που είναι λεχόνες ή έγκυες. Η Προεδρία ε, η Σουηδική Προεδρία έχει, έχει σκοπό να κάνει κάτι και τι περιμένετε από την, Σουηδική, από την Ισπανική συγγνώμη, Προεδρία. Let's, let's start with, Mr. Um, uh, να ξεκινήσουμε τον κύριο Κοφεράτη και το θέμα των μεγαλύτερων σε ηλικία στην αγορά εργασία. Πιστεύω ότι παρότι οι νέοι δεν μπαίνουν στην αγορά εργασία και όλοι ανησυχούμε γι' αυτό, έχουν πολλές ευκαιρίες όταν η οικονομία πάει καλύτερα. Αντίθετα, ένας ηλικιωμένο, ένας άνθρωπος που στο τέλος της διαδρομία του απολύεται, είναι πολύ πιο δύσκολο να ξαναμπεί. Ανησυχώ λοιπόν περισσότερο, ακόμη περισσότερο για τους ηλικιωμένου που μένουν πίσω σε καιρούς κρίσης. Και ένα από τα παραδείγματα που είδαμε και στη Σουηδία και αλλού ήταν ότι υπήρξε μια μόνιμη, ένας μόνιμος αποκλεισμός των ανθρώπων από την αγορά εργασία. Κάποιοι που δεν γύριζαν πίσω ποτέ. Το είχαμε δει και σε προηγούμενες ε, κρίσεις. Και συνεχίζουμε να έχουμε προβλήματα σήμερα, 15-20 χρόνια μετά την, μεγάλη, την τελευταία μεγάλη κρίση. Αυτό το πρόβλημα το είδαμε στη Σουηδία. Από την άλλη πλευρά, Για παράδειγμα, όταν κλείνουν οι βιομηχανίες, ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι και κρίση οικονομική και κρίση επιχειρηματικού κύκλου, αλλά και αλλαγή της οικονομίας, μεταμόρφωση της οικονομίας που συνδέονται. Και δεν είναι εύκολο να πας στη Volvo και τη Saab και να πεις στους αυτοκίνητο που είναι εκεί χρόνια και χρόνια ότι Ο εργαζόμενο στην, στην αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει να πάει ξανά στο σχολείο και να γίνει νοσοκόμο. Χρειάζεται, είναι σύμφωνο ότι χρειάζεται συντονισμό όλων των πολιτικών. Δεν μπορεί να έχουμε τι ε, πολιτικέ ε, θέσει εργασία ω ένα απομονωμένο νησί. Πρέπει να δουλέψουμε σε συνεργασία με την φορολογική, τη βιομηχανική, την εκπαιδευτική πολιτικέ και με όλου του άλλου τομεί για να μπορέσει να υπάρξει ένα το καλύτερο policy mix, το οποίο θα διαφέρει από χώρα σε χώρα. Γιατί έχουμε διαφορετικά προβλήματα. Και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε το σωστό μείγμα εργαλείων. Χωρίς όμως συντονισμό και ένταξη των ε, πολιτικών, χαθήκαμε. Θα είμαστε σαν του ασφαλιστές που πηγαίνουν στο σπίτι με το ατύχημα και δεν θα είμαστε πυροσβέστες πριν τη φωτιά. Τώρα για το αν θα δώσουμε προτεραιότητα στα θέματα απασχόληση, η απάντηση είναι ναι. Προφανώ. Είναι ζωτικό το ζήτημα. Αν δεν το κάνουμε αυτό, να πάμε σπίτια μα. Και ο λόγο είναι απλό. Για να επανέλθω σε αυτά που είπα νωρίτερα. αν δεν έχουμε υγεία αγορά εργασία, θα συζητάμε για το πώ θα ξοδέψουμε χρήματα που δεν θα αποκτήσουμε ποτέ, που δεν θα έχουμε. Πρέπει λοιπόν το θέμα να είναι στην, στην ατζέντα. Κατόπιν. Για τα άλλα θέματα, τι θα γίνει στο μέλλον, τι θα κάνουμε στην μελλοντική. Καλύτερα θα ήταν να μην απαντήσω εγώ, να το απαντήσει ο συνάδελφος ο Ισπανός καλύτερα το ξέρει το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι ο επόμενος επίτροπος θα αντιμετωπίσει πολύ σημαντικά ζητήματα στην ε, Επιτροπή και με την Επιτροπή σας κιόλας και του εύχομαι καλή επιτυχία. Αγωνία λοιπόν για όλους. Ο κύριος Λεβινγκστον και η κυρία Λίζα Καντσαρή. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ να σας βλέπουμε πάντα κοντά μας. Μας δίνει τη δυνατότητα να θέσουμε ερωτήματα. Έχω λοιπόν ερωτήσεις για σας. Αν κατάλαβα καλά τα όσα είπατε, θεωρείτε ότι, ότι δεν ήταν το Λαβάλ μια καλή απόφαση όπως και οι αποφάσεις Viking. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αυτή η οδηγία η οποία οδήγησε σε κάποιες λύσεις μπορούμε να πούμε ότι είναι μινιμαλιστική αυτή η οδηγία. Ξεκίνησε από κάποιες περιπτώσεις και έδωσε μινιμαλιστικές λύσεις. Ωραία. Λοιπόν, και εμείς πρέπει κάτι να κάνουμε ώστε τα συμπεράσματα του δικαστηρίου να εφαρμοστούν. Αλλά σαν πολίτες της Ευρώπης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλοι έχουμε το δικαίωμα να προασπίζουμε την κοινωνική μας και οικονομική μας ευημερία. Ελπίζω λοιπόν ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε ώστε οι διατάξεις που εγκρίθηκαν να εφαρμοστούν κιόλας. Όσον αφορά τώρα την οδηγία για το χρόνο εργασίας που συζητήθηκε μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Η Κομισιόν πέρασε ένα μήνυμα, ανησυχο, ανησυχητικό θα έλεγα, το εξή. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το Ευρωκοινοβούλιο, όπως το ξέρετε και εσείς σίγουρα, επανειλημμένα ζήτησε τη μείωση, την κατάργηση μάλιστα, της ποσόστοσης που μειώνει τις δυνατότητες των μισθωτών να εργαστούν σε, ορισμένες, ορισμένα μέρη. Ποια είναι η άποψή σας λοιπόν, ποια είναι η άποψη δηλαδή της Προεδρίας της Σουηδικής όταν θα φτάσετε να το συζητήσετε αυτό το ζήτημα. Επίσης, Υπουργέ, ξέρετε την έκθεση της ομάδας Στόιμπερ, η οποία αναφέρεται σε ορισμένες ρυθμίσεις για τους μισθωτούς στις μικρομεσαίες. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό διοικητικό βάρος, τεράστιο θα έλεγα για τις μικρομεσαίες, αν τηρηθούν όλες αυτές οι διατάξεις. Ποια είναι η άποψή σας λοιπόν σε σχέση με αυτούς τους κανόνες και τι πιστεύετε για τα συμπεράσματα στο ΙΜΠΕΡ. Τι πρόβλεψη κάνετε κύριε Υπουργέ για το μέλλον. Πιστεύετε ότι είναι σκόπιμο να γίνεται μια εξέρεξη για μεγάλη ομάδα μισθωτών, μια εξαίρεση από τους κανόνες της απασχόλησης και από τους κανόνες του περιβάλλοντος εργασίας. Βεβαίως πρέπει να μειωθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις, αλλά όχι σε βάρος της υγείας των μισθωτών. Θέλω την απάντησή σας. Ακόμη, μιλήσατε για την κοινωνική Ευρώπη. Είπατε ότι η κοινωνική Ευρώπη ξεκινάει με την απασχόληση. Πολύ ωραία ιδέα σας. Συμφωνώ. Θα ήθελα όμως να προσθέσω ότι όταν μιλάμε για απασχόληση πρέπει να μιλάμε για καλές θέσεις εργασίας. Καλές, επαναλαμβάνω, καλές συνθήκες εργασίας, καλό περιβάλλον εργασίας, καλή ασφάλεια. Να λοιπόν ερωτήσει που έχω για σας. Πιστεύω ότι μπορεί να μην συμφωνείτε μαζί μου αλλά τουλάχιστον θα μας πείτε την άποψή σας. Λοιπόν, η δυνατότητα εργασίας είναι, αν θέλετε, η αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πρέπει να τις δώσουμε και ένα θετικό περιεχόμενο. Έχουν υπάρξει καταχρήσεις σε αυτόν τον τομέα που πρέπει να καταπολεμηθούν άμεσα. Σε ορισμένε εταιρείε λοιπόν ε, απολύουν τους μισθωτού του και προσλαμβάνουν από άλλη χώρα. Αυτό είναι η λάθος ερμηνεία της κινητικότητας. Υπάρχει όμως και άλλο πρόβλημα. Η αναγκαστική εργασία. Το εμπόριο ανθρώπων η υποχρεωτική εργασία είναι μεγαλύτερες ε, σήμερα σε διαστάσεις στην Ευρώπη από την εποχή της δουλείας. Λοιπόν, μην το παραμερίζουμε αυτό. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Τι γίνεται μετά από μία κρίση Λοιπόν, μετά από μία κρίση υπάρχει μία μακρά περίοδος έτσι, αδράνειας και στη Φιλανδία και στην Σουηδία θα έχουμε μακρά περίοδο ανεργίας ουσιαστικά και πρέπει να δούμε πόσο μακροπρόθεσμη ανεργία θα υπάρξει. Θα συζητάμε λοιπόν αυτά στη Φιλανδία. Μιλάμε επίσης για τα νέα νομοθετήματα για τον ανταγωνισμό. Έχουμε νομοθετήματα de που επηρεάζουν τον τρίτο τομέα Υπάρχουν δηλαδή αυτοί που έχουν τις δικές τους επιχειρήσεις αλλά απειλούνται εξ αυτής της νομοθεσίας που περιορίζει τις δραστηριότητές τους. Έχετε ευαίσθητα αυτιά κύριε Υπουργέ, είπατε πολύ ωραία. Λοιπόν αναρωτιάμαι αν έχετε ακούσει απόϊχους αυτού του τύπου ως τώρα. Yes, thank you very much. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσω λίγο για την απόφαση Λαβάλ και τις άλλες αποφάσεις που εντωμεταξύ εκδόθηκαν. Βεβαίω δεν μπορώ να κάνω συμπίκνωση των νομικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά βεβαίω ήμασταν πολύ δυσαρεστημένοι. Δεν είναι μυστικό αυτό με την απόφαση. Το θέμα είναι τώρα, μπορούμε να κάνουμε κάτι για να καταπολεμήσουμε αυτή την κατάσταση η ρητορική μου ερώτηση θα ήταν τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Το μόνο που ακούσαμε σαν εφικτό είναι είτε μια κοινωνική ρήτρα συνδεδεμένη με τη συνθήκη και αυτό είναι ξεπερασμένο πια, δεν, είναι εφικτό, ή μία αναθεώρηση της οδηγίας. Αυτά είναι τα δύο πράγματα που έχουν προταθεί κατά τη διάρκεια των όλων συζητήσεων. Έχω θέσει επαναλημμένα το ζήτημα στο Συμβούλιο Μάλιστα στην πρώτη συνεδρίαση μετά από αυτή την δικαστική απόφαση και δεν υπάρχει καμία υποστήριξη στο Συμβούλιο για αναθεώρηση της οδηγίας για την τοποθέτηση των εργαζόμενων. Βεβαίω η μπάλα είναι στο γήπεδο της Κομισιόν. Η Κομισιόν θα ενεργήσει, αν ενεργήσει κάποιος, πρέπει να αποσαφινιστεί μάλιστα ε, το τι σήμαινε ο πρόεδρος, το τι εννοούσε μάλλον με συγχωρείτε, ο πρόεδρος Μπαρόσο όταν μιλούσε για κάποια οδηγία. Βεβαίως είναι σημαντική η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Η Κομισιόν μέχρι τώρα υπήρξε αρκετά αποτελεσματική συνοργάνωση μιας ανταλλαγής πληροφοριών πιο διαφανούς με τα συνδικάτα και τα λοιπά και περιμένω περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες, λεπτομέρειες όσον αφορά την οδηγία τοποθέτηση εργαζόμενων. Αλλά δεν, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι κανείς δεν θέλει την αναθεώρηση στο Συμβούλιο. Τώρα, όσον αφορά την οδηγία για τον χρόνο εργασίας. Θυμόσαστε το σχέδιο με τον πεθαμένο παπαγάλο του Μόντι Πάιθον. Λοιπόν, το Συμβούλιο κατάφερε να φτάσει σε μια συμφωνία μετά από 7 χρόνια και όλα καταστράφησαν όταν ε, μπήκαμε σε διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Όταν λοιπόν συναντηθείτε με τον νέο Επίτροπο, σας παρακαλώ να το ρωτήσετε τι θα κάνει, γιατί δεν έχουμε καμία ιδέα εμείς. Πιστεύω λοιπόν ότι τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες η συζήτηση έχει δημιουργήσει μια νέα κατεύθυνση, έχει ανοίξει μια νέα κατεύθυνση για τον χρόνο εργασίας. Ε, το σκηνικό δηλαδή είναι ενδιαφέρον όσον αφορά τις εξελίξεις τα επόμενα χρόνια. Η θέση της Σουηδίας και η προσωπική μου θέση ήταν να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάποια συμφωνία για την οδηγία χρόνου εργασίας διότι έχουμε με 23 άλλες χώρες τουλάχιστον προβλήματα όσον αφορά την ερμηνεία της σημερινής οδηγίας. Οπωσδήποτε θα θέλαμε η οδηγία χρόνου εργασίας να αφήσει ε, περιθώριο συμφωνίας για τους κοινωνικούς εταίρους. Κατανοούμε ότι η δυνατότητα opt-out είναι περίπλοκο ζήτημα και οι χώρες που έχουν opt-out σήμερα δεν έχουν κανέναν λόγο να έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμφωνήσουν. Μπορούν απλώ να μείνουν σπίτι και να λένε όχι, δεν θέλουμε συμφωνία. Και γι' αυτό χρειάστηκε τόσο χρόνο στο Συμβούλιο και λυπάμαι που δεν προχώρησε και μετά. Τώρα, η ομάδα στο ΟΜΠΙΠ. Αυτό θα το συζητήσουμε και εσωτερικά και διεθνώς. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ χαζή ιδέα να αποκλείσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να γίνει αξιολόγηση του κινδύνου και με βάση τον κίνδυνο και τις πιθανότητες και τις πραγματικές περιπτώσεις να γίνουν οι εξαιρεσει ή να αποκλειστούν ορισμένε περιπτώσεις. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα ενεργήσουμε με βάση την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Πασκάλ Λογκάρη και μετά ο κύριος Ρίτσαρτ Φαρμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ για τις επεξηγήσεις σας και για τις ενέργειές σας. Λοιπόν, το θέμα ουσίας που ελάχιστα συζητάμε εδώ είναι το εξής. Η ενεργεία αυξάνεται και συνεχίζει να αυξάνεται. Αυξήθηκε και αυξάνεται. Είναι λοιπόν το θέμα ουσίας με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε. Να συζητήσουμε δηλαδή τα απαραίτητα μέτρα για να υποσχωρήσει η ανεργία. Τα μέτρα που αναφέρατε είναι σίγουρα ενδιαφέροντα, αλλά δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τη ροή της ανεργίας που οδηγεί σε μεγάλη φτώχεια. Δεύτερον, μου κάνει πολύ εντύπωση η απάντησή σας στην συνάδελφο Τούρινεν όσον αφορά το κοινωνικό dumping και τη μεταφορά εγκαταστάσεων. Δεν είναι οι μισθωτοί που αποφασίζουν να αλλάξουν χώρο για να πάνε να εργαστούν. Οι επιχειρήσεις αλλάζουν χώρο εγκατάστασης, τόπο εγκατάστασης για να υποφεληθούν από τις φορολογικές και κοινωνικές ρυθμίσεις. Επειδή δεν υπάρχει εναρμόνιση Στη Γαλλία έχουμε δύο πρόσφατες περιπτώσεις. Υπάρχει μια επιχείρηση στην Ile de France, μιας, της H&M, μεγάλος όμιλος και κάνει θηγατρική την τροφοδοσία της για να μπορέσει αύριο να μεταφέρει αυτούς που είναι στον μπουρζέ, τους εργαζόμενους, στη σφυδία. Λοιπόν, υπάρχει ακόμη μία άλλη που φτιάχνει Ρουλεμάν, η SKF, η οποία δεν της έφτασε που έκλεισε το εργοστάσιο της στη Βοντέ πρόσφατα, αλλά ζητά από τους μισθωτούς που απέλησε να πάνε να εκπαιδεύσουν τους εργάτες που τους ανταγωνίζονται στη Βουλγαρία. Λοιπόν, είναι αυτό το μοντέλο της κοινωνικής Ευρώπης που αναζητούμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν πρόκειται να υποστηρίξω μια τέτοια Ευρώπη. Τρίτον, αντιλαμβάνομαι το στόχο σας για την κοινωνική συμπερίληψη, αλλά δεν θα υπάρξει τέτοια ένταξη κοινωνική παρά μόνο αν καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες για την έρευνα και για τις πιστώσεις κατάρτισης των αυριανών επαγγελμάτων, διότι πρέπει να επινοηθούν αυριανά επαγγέλματα. επαγγέλματα. Τέταρτον, θα υποστηρίξω τις προτάσεις για τις μικροπιστώσεις αλλά θεωρώ ότι το θέμα των πιστώσεων και του ρόλου της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών για την ύπαρξη χαμηλού ή μηδενικού επιτοκίου στις πιστώσεις που δίνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που καταρτίζουν και προχωρούν είναι ένα ζήτημα πολύ ευρύτερο από ό,τι το διατυπώνουμε. Λοιπόν, η ιδέα του να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ταμείο για την απασχόληση και την κατάρτιση είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορούμε να εξετάσουμε σοβαρά σήμερα για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, πριν από έξι μήνες διατύπωσα εδώ μέσα πόσο απογοητευμένος είμαι εκ του γεγονότος ότι η Προεδρία της Σουηδίας παρουσίασε το πρόγραμμά της. Ήμουν απογοητευμένη δηλαδή, είμαι απογοητευμένος με το πρόγραμμά της. Λοιπόν, οι φόβοι μου απαληθεύτηκαν δυστυχώ. Κατά την άποψή μου η Σουηδική Προεδρία δεν θα γράψει το όνομά της στην ιστορία των Προεδριών με χρυσά γράμματα. Ειδικότερα δε σε αυτό το τομέα που μας απασχολεί. Τα ερωτήματα που ήθελα να σας κάνω τα κάναν άλλοι. Λοιπόν δεν θα τα επαναλάβω. Έχω όμως μια ερώτηση ουσία και θέλω την άποψή σα από αυτό. Ετοιμάζεται μία συμφωνία με την Κολομβία συνθήκη, σύμβαση. Επικρίνεται από τα συνδικάτα με τον ίδιο τρόπο όπως η συμφωνία με την Νότια Κορέα. Η Κολομπία είναι μια χώρα όπου, όπου την ανάληψη της εξουσίας από τον πρόεδρο Ουρίμπε, τον οποίο παρουσιάζανε σαν μεγάλο δημοκράτη, 500 συνδικαλιστές δολοφονήθηκαν. Το να γίνει κανείς ε, επικεφαλής ε, συνδικαλιστής είναι σαν θανατική ποινή ε, και εκτέλεση. Κάποιος τους δολοφονεί συνεχώς. Ποια είναι η άποψή σας λοιπόν σε σχέση με αυτή τη σύμβαση ή συμφωνία που έχει κατά νου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ελεύθερο εμπόριο με την Κολομβία. Thank Θα προσπαθήσω να μιλήσω πρώτα για την SKF και την H&M. Βεβαίως δεν εξουσιοδοτούμε να μιλήσω για αυτές τις περιπτώσεις, ξέρω πολύ λίγα, αλλά νομίζω ότι τα φορολογικά είναι αυτά που κυριαρχούν. Δεν έχει σχέση με την υπόθεση Λαβάλ. Επανέρχομαι όμως στο βασικό ερώτημα. Τι δημιουργεί θέσεις εργασίας. Πρώτον, από την έρευνα και την εμπειρία έχουμε διαπιστώσει ότι η προσφορά είναι μεγάλο ζήτημα. Οδηγεί στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Βεβαίω, αυτό σχετίζεται με τη ζήτηση καταναλωτικών κτλ. Συνεπώς χρειαζόμαστε και τους πελάτες στην οικονομία. Πελάτες που θέλουν προϊόντα, υπηρεσίες και άλλα διάφορα. Άρα θέλουμε μια οικονομία που να έχει εμπιστοσύνη στο μέλλον της. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε δραστήρια, ε, δραστικά με μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης στις βιομηχανικές χώρες. Επίσης το ίδιο ισχύει και για τις τράπεζες και τις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Δεν προσπαθούμε να σώσουμε τις τράπεζες, τους ιδιοκτήτες, αλλά το αίμα της οικονομίας για να προωθήσουμε την εμπιστοσύνη. Κύριε Φάβρα. Λυπάμαι ε, που δεν σας ευχαριστημένος με τη Σουηδική Προεδρία. Αν ήσασταν, θα ανησυχούσα γιατί δεν έχουμε τις ίδιες πολιτικές φιλοδοξίες. Άλλο ζήτημα βέβαια αυτό. Ως προς την Κολομβία. Ε, πρόκειται για αρμοδιότητα πυρήνα της Κομισιόν και δεν μπορώ να παρέμβω, αλλά από τη Σουηδική ε, προσέγγιση είμαστε ο έκτος χορηγός παγκόσμια και είναι υπόθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας να παρακολουθήσει αυτό το ζήτημα. Και δεν είναι αποδεκτό. Η κατάσταση δηλαδή που περιγράψατε είναι απαράδεκτη, συμφωνώ μαζί σας και προσπαθούμε όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε ο ILO να μπορέσει να κάνει ό,τι χρειάζεται σε αυτό το τομέα. Όταν ε, αναφερόμαστε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, όμως θα πρέπει να ζητήσω τη συνδρομή της Κομισιόν για να σας απαντήσει. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, τελευταίος ομιλητής, η κυρία Βερόνικα Λοπέ Φόντανιε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να θέσω ένα ζήτημα ένα ερώτημα το οποίο ήδη έχει τεθεί σε σχέση με τα, ε, τους αναπήρους. Το ΕΛΚ είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί πολύ και φαντάζομαι ότι και άλλες συμμάδες θα θέλουν να ξέρουν ποια, έχει, ποια είναι η κατάσταση με τα ΑΜΕΑ. Έχουν τεράστιες δυσκολίες να βρουν θέσεις εργασίας. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στη δικιά σας τη χώρα, αλλά μπορώ να σας πω ότι στην Ισπανία η δημόσια διοίκηση έχει κάποιο ποσοστό θέσεων για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες, αλλά αυτές οι θέσεις πολύ συχνά μένουν κενές. Άρα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Να εξασφαλίσουμε ένα λογικό μέλλον για αυτά τα άτομα. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία ε, τα οποία θα μπορούσαν να μας ενδιαφέρουν. Ε, η απασχόληση τους έχει θίξει περισσότερο από άλλες ομάδες των πολιτών. Ποια είναι οι μελλοντικέ δυνατότητες. Ευχαριστώ κύριε Λόπες. Μια τελευταία ερώτηση και εγώ υποφελούμαι τις ευκαιρίες κύριε Υπουργέ. Είπατε εισαγωγικά, μάλλον αναφερθήκατε εισαγωγικά και στην θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας και της του ξεκινήματος της διαδικασίας για τη στρατηγική 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως κράτος μέλος, τι περιμένετε από την θέση ισχύ της συνθήκης. Όχι τόσο ως προεδρεύων, αλλά ως κράτος μέλος. Ιδίως στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών. Θεωρείται σημαντικό να χρησιμοποιεί το Συμβούλιο και πώς τις διατάξεις της συνθήκης στον τομέα τον κοινωνικό. Δεύτερον, η στρατηγική 2020, όπως τη λέμε πλέον. Εγώ πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγει από το γεγονός ότι το κολέγιο, το παλαιό κολέγιο που τώρα είναι ένα μονοκέφαλο ζώων μόνο με τον πρόεδρο διαμορφώνει τη στρατηγική της Ένωσης τα επόμενα δέκα χρόνια. Τέλος πάντων, ίσως όμως η Επιτροπή να είναι ένα ζώο πανέξυπνο, έστω και ένα κεφάλι. Για την στρατηγική. Ως ε, Σουηδός υπουργό. τι θα πείτε στους εταίρους και συναδέλφους σας των άλλων κρατών μελών. και ως μέλος μιας κυβέρνησης σχετικά με την θέση των θεμάτων των οποίων είστε αρμόδιος για, την, για το μέλλον. Διότι μέσα στη στρατηγική υπήρχε ο όρος απασχόληση, πλήρης απασχόληση μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται ωστόσο και χωρίς την κρίση δεν νομίζω ότι θα τα καταφέραναμε να δημιουργήσουμε πλήρη και να αυξήσουμε την απασχόληση. Εάν ξεκινούμε μια νέα στρατηγική τώρα, μια συζήτηση για μια νέα στρατηγική, καλύτερα είναι να έχουμε μια εικόνα του που βρισκόμαστε τώρα και να αποφύγουμε να έχουμε ένα, έναν απολογισμό τόσο απογοητευτικό όπως αυτόν τη στρατηγική τη Λισαβόνα. Κάτι άλλο ακόμα. Ποιο είναι κατά την άποψή το χρήσιμο χρονοδιάγραμμα. Και εσείς είστε ειδικό στα θέματα του κοινωνικού διαλόγου, μια και είστε υπουργό απασχόληση τη Σουηδία. Ούτω ώστε οι εταίροι και του κοινωνικού διαλόγου και θεσμικά να μπορέσουν να μετάσχουν ε, αποτελεσματικά στη στρατηγική. Διότι ο σύγχρονο κόσμο τη επικοινωνία μα μαθαίνει ότι για να πετύχει πρέπει να του εμπλέξει όλου. Ένας, ένα ακέφαλο ζώο μπορεί, δεν μπορεί να καθορίζει τις στρατηγικές ο Σουηδός υπουργό. πώς τη βλέπετε την ε, νέα αυτή στρατηγική. Προφανώς αυτό ξεπερνάει την ε, θητεία σας, αλλά επειδή είσαστε και προνομίχους συνομιλητής μας, ε, δεν διστάζω να σας θέσω αυτό το ερώτημα. Να ξεκινήσω με το ερώτημα της κυρίας Λόπε Φοντανία για τα άτομα με αναπηρίες. Δύο θέματα πρέπει να δούμε. Πρώτον, και αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι που παίρνουν ταυτού στην αγορά εργασία. Γι' αυτό στην, στο ξεκίνημα της ε, παρέμβασής μας μίλησε για το άτομο που ήταν σε αναπηρικό καροτσάκι για χρόνια. Προφανώ η κατάσταση των ατόμων με αναπηρίε ποικίλει από κράτο σε κράτο ανάλογα με την κατάσταση. Στη Σουηδία, για να σα δώσω ένα παράδειγμα τη δική μου χώρα, ξοδεύουμε κάθε χρόνο 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε επικουρία, σε βοήθεια των αναπήρων στην αγορά εργασία. Πολλά λεφτά για μια μικρή χώρα. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα συνδυασμό μεθόδων. Ενισχύσει, επιδότηση δηλαδή, βοήθεια για να τύχουν αργής και σε επίπεδο ανθρώπων, διευκόλυνση στο χώρο εργασία, διευκόλυνση του χώρου εργασία, συγγνώμη, για να είναι πιο προσπελάσιμο σε άτομα αναπηρίε. Δουλεύουμε και με νομοθεσία κατά της, ε, των διακρίσεων, με δομέ ε, αναφορών, σε συνεργασία με του κοινωνικού εταίρου. προσπαθώντας να εκπαιδεύσουμε και να παροτρύνουμε τους, προ, τους ε, εργοδότες να προσλαμβάνουν άτομα αναπηρίες. Αλλά παρά τα κονδύλια, όπως σωστά είπατε, η πραγματικότητα είναι ότι σε δις, σε χαλεπούς οικονομικούς καιρούς μειώνεται το ποσοστό εργασίας των ατόμων με αναπηρίες. Και αυτό είναι πραγματικά κρίμα. Χρειαζόμαστε τον καθένα και να σα δώσω παράδειγμα. Έχουμε άτομα που μπορούν και θα έπρεπε να είναι κομμάτια της Ή που χρησιμοποιούμε τους πόρου του κατά κάποιο τρόπο. τι γνώσει και την ανάγκη τους να μπουν στην αγορά εργασία. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν να βελτιωνόμαστε σε ό,τι αφορά την πρόσβαση, το να τους, παραχωρούμε, τους δίνουμε πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Όλα τα κράτη-μέλη το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν με διαφορετικού τρόπου που προσπαθούν να καταπολεμήσουν την απομάκρυνση αυτή από την. Ε, δεν υπάρχει ένα ε, δρόμο. Υπάρχουν ε, νομοθεσίε, παιχνίδια ρόλων, ενισχύσει. Στην ενδιαφέρουσα ερώτηση τη κυρία Μπερέ, εγώ θα έλεγα ότι Προέρχομαι από μια χώρα όπου λέμε ότι έχουμε καλό κοινωνικό διάλογο. Και γι' αυτό θεωρώ καθοριστικό να υπάρξει χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα μετάσχουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές. Ούτως ώστε να υπάρξει, αν όχι 100% συμφωνία για την ε, ατζέντα μετά τη Λισαβόνα, μια υψηλή αποδοχή του τρόπου με τον οποίο θα δουλέψουμε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μία ε, απογοήτευση και με την υφιστάμενη κατάσταση που δεν έχουμε επιτροπή, που δεν έχουμε επιτροπή και θυμίζει λίγο Ξέρετε ότι καμιά φορά που χρειάζεται να αλλάξει, ε, να να αλλάξει κινητήρα του αεροπλάνου, την ώρα πετάει. Εμείς πάντως πιστεύουμε ότι ήταν σημαντικό το Συμβούλιο Απασχόλησης να περάσει ένα σαφές μήνυμα και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δικαιωματικού και στην Ισπανική Προεδρία για τα σημαντικά συμπεράσματα. Δεν ξέρω αν η απάντηση είναι αρκή, αρκετή. Όχι, δεν είναι προφανές. Θα ήταν ίσως καλύτερο. Κανονικά, τα θέματα το, της ατζέντα μετά τη Λισαβόνα θα πρέπει να αντικείμενο τη Συνόδου Κορυφή του Μαρτίου. Το, το κάναμε νωρίτερα. Εγώ πιστεύω ότι ελπίζω η Ισπανική Προεδρία να εμπλέξει όλε τι πλευρέ το στομότερο δυνατό. Και πιστεύω ότι η ένταξη πολιτικών είναι ακριβώ. Δηλαδή να υπάρξει μία σύγκληση όλων των πολιτικών προς την αγορά εργασία. Ούτως ώστε να μην θεωρηθεί ότι μία συγκεκριμένη πολιτική ή μία συγκεκριμένη ομάδα έμεινε στο περιθώριο. Και πάλι δύο λέξεις μου έρχονται στο μυαλό. Εκπαίδευση, ενεργοποίηση. Μόνο έτσι μπορούμε να φέρουμε πίσω τον κόσμο. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είμαστε νησί. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια φορολογικών επενδυτικών μισολογικών μέτρων. Κατόπιν, το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα μέσα είναι μεταγενέστερο θέμα. Καταλαβαίνω η θεσμική απογοήτευση, αλλά εγώ δεν μπορώ να συμβάλλω εδώ. Ελπίζω η Κομισιόν να ξεκινήσει να δουλεύει το συντομότερο δυνατό και να αναλάβει και να συνεχίσει τη διαδικασία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ on Lisbon and Λισαβόνα τώρα και δημόσιες υπηρεσίες. Νομίζω ότι και σε τομέα αυτό θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοπορία η Επιτροπή. Το σημειώνουμε, δεν θα πω τίποτα άλλο. Ωραιότατα. Πείτε στους διαδόχους σας ότι θα τους κυνηγάει το Κοινοβούλιο για το ζήτημα αυτό και ότι προφανώς αυτό θα είναι κομμάτι της κοινωνικής ατζέντα. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, δεν τελειώσαμε. Υπάρχει και συμφωνία για την έκθεση Κούνσου σχετικά με, το με τη μικρο χρηματοδότηση. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία αύριο στην Κορεπέρ. Ελπίζοντας ότι ο λόγος τουλάχιστον η λογική δική μας θα κερδίσει. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν σας έκανα τις ανακοινώσεις γιατί ήθελα να δώσω το λόγο στον Υπουργό. Επανέρχομαι για να σας πενθυμίσω τα εξής. Τα πρακτικά της επίσκεψης κάποιων μελών της Επιτροπής μας στο Μπιλμπάο όπου επισκέφθηκαν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια και την Υγιεινή στον χώρο εργασία διανεμήθηκαν στα μέλη. Επίσης, μία αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας πήγε στην Ισπανία 12-13 Νοεμβρίου. Νοεμβρίου. Τα πρακτικά και της επίσκεψης αυτής σας δόθηκαν. Να υπογραμμίσω ότι στη συζήτηση αυτή με την επερχόμενη Προεδρία που θα τη δούμε και τον Ιανουάριο στις συζητήσεις εμφανίστηκε μια σειρά σημαντικών θεμάτων για τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε. Αναφέραμε το ζήτημα της, του χρονοδιαγράμματος για την υιοθέτηση της στρατηγικής 2020. Η ανταλλαγή ήταν χρήσιμη γιατί έδειχνε ότι είναι δύσκολη, ότι ενδεχόμενα είναι δύσκολη η έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο. Να πω επίσης και δύο-τρία πράγματα που τονίστηκαν και που μπορεί να είναι χρήσιμα να έχουμε στο μυαλό μας. Την πρωτοβουλία που θα αναλάβει η Ισπανική Προεδρία για τις δυσκολίες δουλειάς για σχετικά με τους α, ε, ανεξάρτητους εργαζόμενους, ιδιαίτερα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, σε μια χώρα όπου προφανώς ένα μεγάλο τμήμα της παραγωγής είναι στα χέρια των μισθωτών εργαζομένων. αλλά αυτοί οι, οι ανεξάρτητοι δεν έχουν πολλές προστασίες, πολλή δυνατότητα προστασίας. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να μας ενδιαφέρει δώσαμε έμφαση στα ζητήματα μη διάκρισης, συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασία, που και αυτό μπορεί να ενδιαφέρει τα μέλη της Επιτροπής, έγιναν και πολλές συζητήσεις για τα θέματα αγοράς εργασίας και την μη ανάκαμψη της πιστοτικής δραστηριότητας από πλευράς τραπεζών ενώ εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με το τι σημαίνει αυτό για την αγορά εργασία. Αυτά είναι τα κύρια θέματα που πρέπει να κρατήσουμε νομίζω από την επίσκεψη αυτή. Σας καλώ να δείτε τα πρακτικά που σας ανακοινώσαμε. Τελευταίο σημείο. Χρήση του πόρου προσαρμογής ε, των κονδυλίων προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. στι περιπτώσει των εργαζομένων ε, Ολλανδίας, Αυστρίας και Σουηδίας, ε, για του οποίου ξεκίνησε από μας, ε, έγινε η προσφυγή σε εμά, ξεκίνησε μια ομάδα εργασία που ενέκριναν οι συντονιστέ και μεταβιβάστηκαν στον εισηγητή του, του, του, της Επιτροπής Προλογισμού, κύριο Μπέγκ. Αυτά για τις ανακοινώσεις. Να σας τονίσω ότι έχουμε τρεις νέους φοιτητές μεταξύ μας που κάνουν μάστερ επαγγέλματα επαγγελμάτων Ευρώπης από τη Σορβόνη. Καλώς ήλθατε στις εργασίες μας. Σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Όπως συμφωνήσαμε, Επειδή λείπει η εισηγήτρια θα κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων γιατί στο πολιχείτη στις 26 Ιανουαρίου, δεύτερη συνάντηση, θα γίνει συζήτηση παρούσης και της ηγήτρες. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε την επόμενη 27 μια και η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, επιτροπή γυναικών δηλαδή έχει θέσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πιστεύω ότι θα έπρεπε πριν κάνουμε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων που θα δείξει τις προτεραιότητες και την άποψη που έχουν ε, οι ομάδες για να ενημερώσουμε σχετικά την εισηγήτρια και να της επιτρέψουμε να δουλέψει με τις απόψεις των μεν και των δε. Είπαμε λείπει η κυρία Ροβάνα Πλάμπ και πιστεύω ότι ο κύριος Λίβινγκστον θα μιλήσει εξ ονοματός Παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε. Είπαμε ότι θα κατεγράφονται όλα αυτά που αναφέρονται και θα αποσταλούν απλώς στην εισηγήτρια, τίποτα άλλο. Merci beaucoup. Euh, Madame Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρονή. Ευχαριστώ. Κρίμα που λείπει η συγκήτρια. Ε, πραγματικά με απογοητεύει αυτό. Και πραγματικά είναι δύσκολο να προχωρήσουμε στις δουλειές μας. Να σας πω ότι η οδηγία ήταν για τις γυναίκες καταρχήν. Άρα, ό,τι αφορούσε τους άνδρες, Μπορεί να το συζητήσουμε στο μέλλον, αλλά οι τροπολογίε είναι τροπολογίες οι οποίες έχουν, δηλαδή οι τροπολογίες που μιλούν ε, για άδεια πατρότητα ενώ ακόμα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει την αδιαμητρότητα, είναι κάπως πρόημο. Τα δικαιώματα ανδρών και γυναικών δεν είναι στο ίδιο επίπεδο σε άλλου τομείς. Τώρα, για την περίοδο άδεια μητρότητα. Η διάρκεια των 18 εβδομάδων για μα είναι κάτι το ισορροπημένο που δεν εμποδίζει την δουλειά των γυναικών αλλά ταυτόχρονα πιστεύω βελτιώνει την κατάσταση στα περισσότερα κράτη-μέλη. Το δικαίωμα ελεύθερη γυναίκας που έχουν οι γυναίκες για το πότε θα το βάλουν, πότε το πάρουν, πότε θα βάλουν αυτή την άδεια μέχρι την γέννηση, μέχρι τη γέννηση δηλαδή, μέχρι τον τοκετό είναι κάτι θετικό και πιστεύω ότι αυτή την ελευθερία επιλογή πρέπει να την αφήσουμε. Οι τροπολογίε που μιλούν για την άδεια του πατέρα, επαναλαμβάνω δεν, δεν είναι θέμα κατά την άποψή μου, άλλη είναι η οδηγία, μίλησε και ο Σουηδό υπουργό για μια μελλοντική οδηγία. Σε άλλους τομεί πρέπει να μπουν λοιπόν τα θέματα της άδεια πατρότητας. Αμοιβή κατά τη διάρκεια της άδεια μητρότητας. Εγώ υποστήριζω την πρόταση τη Κομισιόν που προβλέπει και αναφέρεται στην αρχή της επικουρικότητας, προβλέπει ωστόσο η Επιτροπή το δικαίωμα πλήρους εισπρατώμενου μισθού, δεν είναι δεσμευτικό ωστόσο αυτό, αλλά το ποσό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από αυτό της, του επιδόματος ασθένειας. Εγώ το θεωρώ θετικό αυτό. Η πληρωμή στο ακέραιο ε, θέτει ερωτήματα του ποιος θα τα πληρώσει. Η ε, ασφαλιστικοί φορείς, ε, ο εργοδότης, πιστεύω ότι δεν πρέπει να έχουμε δεσμευτική παρουσία εδώ, αλλά να αφήσουμε στα κράτη-μέλη την τελική επιλογή. Για την περίοδο προειδοποίησης τρεις μήνες πριν την άδεια μητρότητας είναι κάτι το θετικό. Η ένταξη των ανεξαρτήτων στην οδηγία πρέπει να το αφήσουμε σε μια άλλη οδηγία που θα διευκρινίζει την κατάσταση των ανεξαρτήτων εργαζομένων σε άλλους τομείς και να αντιμετωπίσει και το θέμα των εγγύων ανεξαρτήτων γυναικών. Για τον, τους πρόορους τοκετούς και τις συνέπειες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Πιστεύω ότι και εδώ πρέπει να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη. Για την αναγνώριση τη ε, μετά, το, ε, τον τοκετό κατάθλιψης ε, δεν νομίζω ότι κατάθλιψης, συγγνώμη, δεν νομίζω ότι είναι θέμα που μπαίνει σε ζητήματα άδεια μητρότητα, αλλά είναι καθαρά ιατρικό ζήτημα και εκεί πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Για την λήψη υπόψη της ε, άδεια μητρότητα σαν, συνταξιοδοτική, σαν περίοδο συνταξιοδότησης είναι κάτι πολύ σημαντικό και ουσιαστικό να θεωρηθεί ότι είναι πραγματική, πραγματικά ε, παρασχεθής εργασία. Για την περίοδο γαλούχησης η χρησιμοποίηση άδεια αυτή κατά την περίοδο των δύο ετών γαλούχησης είναι μια επιλογή τη γυναίκα. Κάποιε κάποιες ε, δεν μπορούν να φυλάσουν κατά συνέπεια δεν πρέπει να τις στιγματίζουμε αυτές αλλά πρέπει να προκρατηθεί και για αυτές τις περιόδους των δύο ετών για τις παρένθετες μητέρες την, ε, είναι ένα ζήτημα πολύ δύσκολο που πρέπει να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη περίπτωση Εγώ είμαι υπέρ από την άλλη πλευρά μια σειρά συμπληρωματικών ε, προϋποθέσεων για τις μητέρες ε, ατόμων με αναπηρίες ή για, τις πολλαπλές, για, για, τους πολλαπλούς, για, τις για τα, πολυ, τα πολύδημα, δίδυμα και παραπάνω. Αυτά. Merci beaucoup. Euh, Madame Cornelissen. Ευχαριστώ. Η κυρία Κορνέλισεν. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε την έκθεση αυτή στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών. Ευτυχώς η κυρία Πλαμή ήταν εκεί το πρωί, οπότε ακούσαμε και τη δική της άποψη. Η ομάδα των Πρασίνων υποστηρίζει την κυρία Στρέλα και τη γραμμή που έχει ακολουθήσει για την ε, έκθεσή της. Ελπίζω ότι η γνωμοδότηση θα, που θα δοθεί ε, θα υποστηρίζει και τη γραμμή της κυρίας Εστρέλα. Δύο πράγματα θεωρούμε οι πράσινοι ότι είναι πολύ σημαντικά. Καταρχήν, η διάρκεια της άδειας μητρότητας πρέπει να αυξηθεί εμείς θέλαμε να πάει στις 24 εβδομάδες. Είναι η μόνη περίοδος που μπορεί να είναι αντικειμενική. Η ΠΟΗ συστήνει τις 24 εβδομάδες γιατί συμπίπτει με τους 6 μήνες κατά τους οποίους πρέπει οι μητέρες να θυλάζουν τα μωρά τους. Αυτό λοιπόν προτείναμε εμείς να αλλάξει, να τροποποιηθεί. Κάτι άλλο τώρα. Οι δύο εβδομάδες άδεια πατρότητας. Το θέμα δεν είναι απλώς θέμα υγείας για την, θέμα, αυτή οδηγία, αλλά είναι και θέμα ε, σωστής κατανομής ε, των βαρών ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών. ειδικά σε αυτές τις πρώτες εβδομάδες μετά την γέννηση, ως νέος γονιός κάποιος μαθαίνει καταρχήν να αλλάζει τις πάνες του παιδιού του, μαθαίνει να απαντά στο κλάμα του μωρού του, μαθαίνει να φροντίζει το παιδί του. Αν το κάνει κανείς αυτό μόνος του, αν το κάνει αυτό μόνο μια μητέρα, μόνη μια μητέρα, ξεκινά δημιουργώντας έτσι μια τάση που θα είναι και τελικά αυτή που θα ακολουθήσει. Δηλαδή η μητέρα θα αναλάβει ας πούμε την φροντίδα του μωρού και ο, πατέρας μένει λίγο εκτός. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτές τις ε, εβδομάδες όλα αυτά να γίνονται από κοινού με τη μητέρα και τον πατέρα ώστε να υπάρχει σαφής κατανομή της φροντίδας του μωρού. Κάποιες τροπολογίες από το ΕΛΚ τώρα μας με έχουν εκπλήξει. Έλεγε μία ότι η μακρύτερη, περίοδος, η μακρύτερη άδεια περιορίζει τις πιθανότητες επιστροφής της μητέρας. Δηλαδή οι χώρες που έχουν μεγαλύτερη άδεια μητρότητας θα έπρεπε να έχουν υψηλότερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει όμως, οπότε καλύτερα να το ελέγξουμε αυτό. Και κάτι άλλο. Η άδεια, η μεγαλύτερη άδεια, εν από, το, από τη συνηθισμένη, δεν χρειάζεται, που, και, που δεν έχει να κάνει με την υγεία της μητέρας. Έχει όμως να κάνει με την υγεία του παιδιού και έχει να κάνει και με το χρόνο που χρειάζεται κανείς για να θυλάσει ένα μωρό. Γιατί εντάξει αυτό μπορεί να το επιλέξει η μητέρα, κανένας δεν μπορεί να της επιβάλλει να θυλάσει το μωρό της. Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο απ' όλα ήταν η τροπολογία για την ε, αναρωτική άδεια. Αν η αναρωτική, αν πρέπει κανείς να λάβει αναρωτική, μια έγκυος γυναίκα, ας πούμε, για πάνω από 6, εβδομάδες πριν τον τοκετό, αυτή η άδεια πρέπει να αφαιρεθεί από την άδεια μητρότητας. Αν δηλαδή μια γυναίκα για δύο εβδομάδες μπει στο νοσοκομείο και μόλις ε, και όταν γεννήσει πρέπει δηλαδή να γυρίσει στη δουλειά δύο εβδομάδες νωρίτερα επειδή πήρε δύο εβδομάδες αναρωτική ε, αυτή η ε, οδηγία γίνεται για να βοηθήσει τις γυναίκες, τις μητέρες, να βοηθήσει τις ε, ε, οικογένειες να κάνουν σωστή κατανομή των βαρών, να βοηθήσει τις γυναίκες να συνδυάσουν την προσωπική ζωή και την επαγγελματική τους ζωή. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Φιγκερέντο με την άδειά σα, γιατί πρέπει να φύγει. Και μετά στον κύριο Πουπάκη. Κύριε Φιγκερέντο. Ευχαριστώ. Και εγώ θα είμαι σύντομη. Όπως αναφέρθηκε η συζήτηση αυτή, έχει ξαναγίνει και στην Επιτροπή Γυναικών και εδώ. Είναι γνωστή και η θέση μας τη ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτική Αριστερά. Υποστηρίζουμε την έκθεση Στρέλα ήδη από την προηγούμενη θητεία και έχουμε την ίδια θέση και τώρα. Θέλουμε βέβαια να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε κάποιες πτυχές που αναφέρθηκαν εδώ και που περιλαμβάνονται στις προτάσεις που έχουμε κάνει. Στι τροπολογίε. Τρία είναι τα βασικά θέματα. Δικαιώματα για τις γυναίκες μητέρες σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει και για τους πατέρες άδεια πατρότητας. Μόνο έτσι θα υπάρξει πραγματικά μοίρασμα των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων της πατρότητας και της μητρότητας και μόνο έτσι οι γυναίκες πέραν του χρόνου που για λόγους υγείας ή άλλους θα χρειαστούν για να αποκατασταθούν θα μπορεί το παιδί να παραμείνει στην ευθύνη και των δύο γονέων προς όφελος και των πατεράδων και των μητέρων και κυρίως των παιδιών των ίδιων να μπορούν και οι δύο να έχουν ευθύνε στον τομέα αυτό. Δεύτερον, όταν μιλούσαμε για δημογραφικά θέματα, είχαμε τονίσει την ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των γεννήσεων, η γονιμότητα. Άρα, να αυξηθεί η αύξηση των αδειών είναι θετική. Και ποτέ, παρόλα αυτά ποτέ ε, σε πολλές χώρες ποτέ η άδεια δεν ήταν ε, ε, ισοδύναμη με τον μισθό. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι υπερβολικό να ζητήσουμε οι άδειε να αμείβονται 100% στον πραγματικό μισθό. Εν τέλει, θεωρούμε να, αναγκαίο να προχωρήσει ταχύτερα η οδηγία, βελτιώνοντας την κατάσταση για το μέλλον. Το ΕΛΚ θα έπρεπε να ξαναδεί τις θέσεις στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Πουπάκη που δέχθηκε να μιλήσει πρώτα η κυρία Φιγκερέδο. Κύριε Πουπάκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε στην πράξη την προσπάθεια που γίνεται για τη συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Είναι επιβεβλημένο να τονώσουμε τη γενετικότητα στην Ευρώπη, σε μια Ευρώπη που γυρνάει ολοένα και περισσότερο, αυξάνοντα παράλληλα τη γενική απασχόληση ώστε να αντιμετωπιστούν σημαντικά θέματα τόσο οικονομικής βιωσιμότητας όσο και γενικού χαρακτήρα. Κατέθεσα κάποιες τροπολογίες σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 9285 που κυρίως έχουν να κάνουν με τη διασφάλιση ελάχιστης υποχρεωτικής άδεια πρώτου και του, τη θεσμοθέτηση ουσιαστικότερης συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων, τη θέσπιση ευέλικτου ωραρίου εργασία κατά διάρκεια γαλουχία χωρί οικονομικέ επιπτώσει για την εργαζόμενη. Πιο συγκεκριμένα, η θεσμοθέτηση ενό ελάχιστου διαστήματο υποχρεωτική άδεια πριν από το τοκετό είναι απαραίτητη σύμφωνα με σχετικέ ιατρικές μελέτε έχουν να κάνουν με την υγεία του μωρού, καθώς με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορεί καμία εργαζόμενη να εξαναγκαστεί να εργαστεί ως το τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης την τελευταία μέρα της. Επιπλέον, οι οικονομικέ διατάξει παρούσας οδηγίας πρέπει να είναι εναρμονισμένες στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων για την ίση μεταχείριση και να ενισχύουν την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων μητέρων. Ακόμα, μέσα σε μια σχέση εργασίας που είναι εκ του προημίου αφοτεροβαρή, το βάρος απόδειξης πρέπει να εναπόκειται σε κάθε περίπτωση στον εργοδότη. Σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά αποδυναμώνεται η θέση της εγγύου εργαζόμενης να διεκδικήσει τα δικαιώματα και την προστασία που της παρέχουν οι διατάξεις της ελληνική Και τέλος, είναι αναγκαία η θέσπιση της επέκτασης προστασίας έναντι αντιπίνων και στους μάρτυρες. καθώ έτσι δίνεται να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και έγκαιρη συμμετοχή του στην εκδίκαση τη καταγγελία, δίχω το φόβο τυχόν δυσμενού μεταχείριση. Η αντίστοιχη τροπολογία είναι σύμφωνη άλλωστε και με τι διατάξει τη οδηγία RECAST 2006-54. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. κύριε Μπάουερ. Ευχαριστώ. Πέρα από το γεγονός ότι αυτό το θέμα Το συζητούμε γιατί είναι σημαντικό. Η έκθεση αυτή έχει πολύ σημαντικά στοιχεία και οι τροπολογίες επίσης. Υπάρχουν όμως κάποια στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο τομέα της ασφάλειας των θέσεων εργασίας. Θα επικεντρωθώ σε κάποια σημεία γιατί θεωρώ ότι αυτά είναι τα πιο συζητη... πολυσυζητημένα στην έκθεση και μπορεί ίσως να δημιουργήσουν προβλήματα μακροπρόθεσμα γιατί είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. Η Επιτροπή λέει ότι αυτή η πρόταση με τον τρόπο που έχει παρουσιαστεί θα είναι αδύνατον να εφαρμοστεί. Αφήστε με να κάνω κάποια σχόλια. Η γονική άδεια που αφορά τους, ε, τους πατέρες, η άδεια πατρότητας. Έχουν γίνει τροποποιήσεις εδώ ως προς αυτό, αλλά θεωρώ ότι η άδεια πατρότητας δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την οδηγία θα ήταν μάλλον καλύτερο να περιμένουμε την Επιτροπή να υποβάλει νέα οδηγία. Και επίσης η γονική άδεια είναι αντικείμενο συζήτηση διαφόρων φορέων. Οι κοινωνικοί εταίροι το συζητούν τώρα, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό να συμπεριληφθεί εδώ. Τροπολογία 41 είναι αδύνατο να την υποστηρίξουμε, πιστεύω. Δεν μπορώ δηλαδή να φανταστώ μια κατάσταση όπου ο εργαζόμενο, ο εργοδότη, συγγνώμη, μπορεί να αξιολογήσει ε, το κίνδυνο που θα έθετε να αμφιβόλω τις δυνατότητες που έχουν οι ε, εργαζόμενοι ή οι εργαζόμενες να τεκνοποιήσουν. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε το σωστό μήνυμα προς τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν ειδικά ε, Ινστιτούτα, ειδικού φορείς ε, για να φροντίζουν τα, τα μωρά. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να μπει σε αυτή την οδηγία. Το βάρος απόδειξης τώρα νομίζω ότι πρέπει να το, ε, από, να το αφαιρέσουμε από την ε, οδηγία. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει. Η οδηγία θα πρέπει να, είναι, να μπορεί να εφαρμοστεί και σε ό,τι αφορά την επιστροφή στην αγορά εργασία. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Madame Nadia Η κυρία Νάντια, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω κι εγώ κάτι για, για την άδεια πατρότητας, η οποία συζητιέται τώρα. Ούτε εγώ ξέρω αν είναι το σωστό σημείο εδώ να τα συμπεριλάβουμε, αλλά σε ό,τι, εν περιπτώσει, ότι είναι, είναι σημαντικό, αν, ε, αν τη συμπεριλάβουμε θα πρέπει να είναι επιπλέον, ε, και να θεωρείται ως επιπλέον άδεια και να είναι εθελούσια. Ε, Επίση μιλούμε για την ε, υγειονομική περίθαλψη της μητέρας μετά, την, ε, μετά τον τοκετό. Συμφωνώ με τις συναδέλφους που λένε ότι θα πρέπει να δώσουμε και στους πατέρες τη δυνατότητα να φροντίζουν από κοινού τις, το παιδί τους με τις μητέρες μητέρες. Αλλά αν αυτό γίνεται θα πρέπει να γίνεται σε ε, εθελούσια βάση. Τώρα, οι υπόλοιπε τροπολογίε που έχουν να κάνουν με διάφορε ειδικέ ε, διατάξει για τα παιδιά με αναπηρία, με, τις, ε, με του πρόρωστοκετού, νομίζω ότι καλό θα ήταν αυτό να το κανονίσουν τα κράτη-μέλη, να το ρυθμίσουν από μόνα του. Ξέρουν επί τόπου ποια είναι η υποδομή που έχουν και μπορούν αυτές οι μεμονωμένε περιπτώσεις να τις υποστηρίξουν. Οπότε νομίζω ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά που σε αυτές τι μεμονωμένε περιπτώσεις πρέπει να ε, εξεύρουν δικέ τους διατάξεις. Για την ευελιξία τώρα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι είναι, υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα, οπότε μια, σε κάποια μπορεί μια γυναίκα να πάρει, ε, να πάρει άδεια λίγο περισσότερη, λίγο λιγότερη, ανάλογα με την εργασία της, πριν τον τογητό, μετά τον τογητό. Εγώ θέλω να έχουμε το δυνατόν περισσότερες επιλογές για τη γυναίκα, να έχει δυνατότητες να διαλέξει με, το, με, με μεγάλο εύρος και αυτές οι έξι εβδομάδες είναι σημαντικές ε, να τις διατηρήσουμε, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να ε, ε, εξεύρουμε εδώ μία διάταξη για όλους, γιατί οι καταστάσει είναι τελείως διαφορετικέ στα κράτη-μέλη. Τώρα, πόσο καιρό θα είναι αυτή η άδεια. Ακούσαμε 14 εβδομάδες, 16, 18, ακούσαμε μέχρι 24 εβδομάδε Ε, εξαρτάται από τη γυναίκα. Αυτό που πρέπει όμως να εγγυηθούμε, να εξασφαλίσουμε, είναι να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι συνθήκες, γιατί κάποιες γυναίκες αντιμετωπίζουν διαφορετικά ε, προβλήματα και είμαστε 20 χρόνια μετά, δεν είμαστε το 1980 τώρα. Υπάρχουν γυναίκε που έχουν την οικογένειά του ε, κοντά του τι βοηθά, τους βοηθά στην, ε, ε, στο να φροντίσουν το παιδί του. Υπάρχουν γυναίκε που δεν βρίσκονται κοντά στην οικογένειά του, που δεν έχουν τη μητέρα του μαζί και είναι μεγάλη πρόκληση να μεγαλώσει μία μάνα το παιδί της από μόνη της. Οπότε νομίζω ότι μια διεύρυνση τη απο μονη τη. οποτε είναι τη αδεια ειναι καλη Οι 18 εβδομάδε ίσω να είναι μια καλή λύση. Παρ' όλα αυτά, ανεξάρτητα από το χρόνο τη άδεια, πιο σημαντικό τη διάρκεια τη άδεια. πιο σημαντικό είναι η αποζημίωση. Η Κομισιόν εδώ και στην πρότασή τη λέει η αποζημίωση 100% του μισθού. Και ελάχιστος μισθό σε περίπτωση ασθένειας. Ε, πρέπει εδώ να έχουμε ένα εύρο όμω, ώστε να μπορεί το κράτο μέλο να κινηθεί μέσα σε αυτό. Έχουμε όμω μια τροπολογία εδώ από τους συντηρητικούς του κυρίου Κάστλερ, την 86, που λέει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θέσουν ένα δικό τους ανώτατο όριο. Και θα ήθελα εδώ να σας προειδοποιήσω να ξεκινούμε τώρα για τις ε, μητέρες να θέτουμε όρια ε, δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Μια γυναίκα όταν έχει γονική άδεια δεν μπορεί να, έχει, να την χάνει διαφορετική μεταχείριση από μια γυναίκα που είναι άρρωστη. Ένα, μια τέτοια, λοιπόν, ένα τέτοιο αίτημα εδώ, να μιλούμε για 76% του μισθού, νομίζω ότι είναι λάθος μήνυμα που δίνουμε στις γυναίκες και είναι και ε, διακριτική μεταχείριση. Ήδη οι γυναίκε ε, λαμβάνουν πολύ, πολύ λιγότερο ε, και πληρώνονται πολύ χειρότερα από τους άντρες Α μην μειώσουμε αυτό ακόμη περισσότερο. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να το αφήσουμε αυτό στα κράτη-μέλη. Δεν μπορούν δηλαδή τα κράτη-μέλη να, να, να δίνουν στην γυναίκα που έχει άδεια μικρότερο μισθό από αυτή που είναι άρρωστη. Εγώ προτιμώ μια γυναίκα να παίρνει άδεια 18 εβδομάδε και να έχει 100% το μισθό τη, παρά να έχει 24 εβδομάδε άδεια και να παίρνει 67% του μισθό τη. Πρέπει λοιπόν να δούμε και βέβαια τι μπορούμε να πάρουμε από όλα αυτά στο από το Συμβούλιο με τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόμας Μαν και μετά ο κύριος Σέρτζιο Κοφεράτη, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με την συνάδελφο, ειδικά για το ότι πρέπει να έχουμε ρυθμίσει στα κράτη-μέλη. Η, ε, αρχή της επικουρικότητας πρέπει να τηρηθεί. Χρειαζόμαστε αρκετές ρυθμίσεις οι οποίες να είναι εθελούσιες. Κάποιες μπορούμε να τις επιβάλλουμε. Ευτυχώς τα πράγματα έχουν αλλάξει. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες μπορούν να διαχειριστούν την κατάστασή τους ε, πολύ καλύτερα, ε, είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένες και μπορούν να φέρουν και τους άντρες πιο κοντά και να τους ε, βοηθήσουν να συμμετάσχουν περισσότερο. Συμφωνώ με την συνάδελφο Μπάουερ, δεν μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε κάπου εκεί να βάλουμε και να ξεχάσουμε και σε μια γωνίτσα την, την άδεια πατρότητας. όταν, είναι, όταν είμαστε σαφεί στου κανόνε μα, τόσο πιο αποδεκτοί θα γίνονται και αυτοί. Η, Σουηδία, το, η Σουηδική Προεδρία το έδωσε μια γραμμή για, τις, για την αγωνική άδεια. Τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό να συμπεριλάβουμε ε, όλα αυτά τα στοιχεία εδώ, γιατί δεν μπορούμε να τα παρουσιάσουμε και στους πολίτες. Τα βάζουμε όλα και εμείς με μια οδηγία και ε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να, να εφαρμοστεί. Σε κάποιους τομείς ε, δεν είμαστε πολύ μακριά από τον άλλον. Ας πούμε, αν δείτε την 52, λέμε ότι χρειάζεται ε, να είναι απρόσκοπτη η επιστροφή της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Και βέβαια πρέπει να δημιουργηθούν και, ε, και ε, οι δομέ πρόνοια για τα μωρά για να μπορέσουν οι γυναίκε να επιστρέψουν στην αγορά εργασία. Πρέπει να υπάρχουν λοιπόν παιδικοί σταθμοί που να μπορούν να πληρωθούν. Ε, σε πολλέ χώρε δεν υπάρχουν τέτοιε εγκαταστάσει, οπότε αυτό είναι ε, αποτρεπτικό για τη γυναίκα. Και δεύτερον πρέπει να μπορούμε ε, να πετύχουμε το, να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση στην αγορά εργασία για τι γυναίκε που επιστρέφουν. Φυσικά υπάρχουν διαφορέ. η κυρία Μπάουερ το είπε. Ε, υγεία και ασφάλεια στην αγορά εργασία. Φυσικά αυτό είναι δική μα αρμοδιότητα. Αλλά άμα αρχίζουμε να διευρύνουμε συνέχεια το πεδίο, ε, δεν θα τα καταφέρουμε καθόλου. Για παράδειγμα, στην 106 του συναδέλφου κάσλερ να πούμε ότι αυτό δεν θα εφαρμόζεται για τις, ανεξα... για τις, ε, για τις ελεύθερες επαγγελματίε. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ε, επικουρικότητα τώρα που πρέπει να τη διατηρήσουμε. Σε πολλές τροπολογίες προσπάθησα να την ε, πω, στην 116, στην 123 και ρωτώ με βάση και την εμπειρία των κρατών μελών. Όντως υπάρχουν, ε, ε, ε εγκαταστάσεις που δεν επιβαρύνονται ιδιαίτερως, που δεν έχουν τόσο πολλή δουλειά Και αν πρέπει να τους επιβάλλουμε νέα καθήκοντα, ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να τους δώσουμε και τις απαραίτητες υποδομές ως προς αυτό. Επομένως πρέπει να τους δώσουμε και την απαραίτητη χρηματοδότηση αυτό. Πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Επίσης είναι σημαντικό να πούμε ότι πρέπει να υπάρξουν αριθμιστικές διατάξεις, ότι στα κράτη-μέλη δηλαδή μπορεί να είναι εφικτά όλα αυτά και ότι επίσης θα, υπάρχει, ε, θα, υπάρχουν, ε, θα υπάρχει ε, χρήση της εμπειρίας των κοινωνικών εταίρων δεν μπορούμε μόνο σε δευτερεύουσες προτάσεις να τα βάζουμε αυτά. Νομίζω ότι ε, υπονομεύουμε το ίδιο μας το έργο. Ε, έχουμε χρόνο να κάνουμε διάλογο, να διαπραγματευτούμε, να κάνουμε και τριμερή διάλογο αν θέλετε, έτσι ώστε να συγκλίνουν λίγο περισσότερο οι θέσεις μας. Να πούμε ότι τώρα αναγνωρίζουμε τι υπάρχει στις, ε, στις τροπολογίες να συνεννοηθούμε τι θέλει ο καθένα. Πολλές φορές μπορούμε ο ένα να εξηγήσει τον άλλον τη θέση του, αλλά οι λεπτομέρειε είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Οπότε ε, ας, έχουμε όλη καλή διάθεση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό μεταξύ των διαφόρων ομάδων. Ο κύριος Κοφεράτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξει προγενέστερη οδηγία. Μεταξύ άλλων και διότι ο κόσμος γύρω μας κινήθηκε ταχύτερα από εμά τους νομοθέτες. Μία νέα διάταξη μπορεί να αφορά κατά απόψή μου δύο βασικά ζητήματα από αυτά που αναφέρθηκαν και αυτά που σχολίασαν οι συνάδελφοι με τροπολογίες. Πρώτον, την παράταση της άδεια, την αμοιβόμενη παράταση. Κάπου, κάποιοι αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο θα αποθάρρυνε την απασχόληση των γυναικών γιατί θα επιβάλλει το κόστος της επιχείρησης. Δεν σημαίνει πουθενά σε καμία χώρα. Δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της διάρκειας άδειας μητρότητας, της αμοιβή τη και της, της πορείας της απασχόλησης των γυναικών. Στη χώρα μου που έχουμε επαρκώς προηγμένους κανόνες ευτυχώς είναι η χώρα όπου η απασχόληση των γυναικών είναι υψηλότερη ποσοστία και εφαρμόζεται η νομοθεσία χωρίς εμπόδια. Αν υπάρχει συνέπεια λοιπόν, συνέπεια ανάποδη είναι ότι αν, έχεις αν δίνεις μεγάλη γονική άδεια, ενθαρρύνεις την ε, γυναικεία απασχόληση. Αλλά σε συζητήσει με τον Υπουργό Εργασία τη Σουηδία χτε, τονίσαμε πόσο σημαντικό είναι να ενθαρρύνουμε την επέκταση και διεύρυνση τη αγορά εργασία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν από τη μια μεριά υπάρχουν διατάξει που έχουν στόχο να προσφέρουν ισότητα ευκαιριών στις γυναίκες όταν η κατάστασή τη είναι χειρότερη και απ' την άλλη να μην νιώμαστε δικαιώματα στους άνδρες. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι το δεύτερο χαρακτηριστικό στοιχείο της διάταξης μπορεί και πρέπει να είναι η άδεια πατρότητας. Δεν είναι, δεν είναι μια αρρύθμιση που θα πρέπει να ενταχθεί αλλού και δεν με πείθει το ότι πρέπει να υπάρχει μια οδηγία για την γονική διάσταση που θα μιλά για την σχέση του μπαμπά με το μωρό. Δεν μιλάμε για την γονική άδεια στο μακροχρόνιο πλαίσιο της ζωής των παιδιών, αλλά για τους πρώτους μήνες της ζωής του νεογνού. Όλοι οι παιδίατροι, όλοι οι ψυχολόγοι μπορεί να σε εξηγήσουν ε, ξεκάθαρα, αυτό είναι δεδομένο πλέον, ότι είναι πολύ σημαντικό το μωρό να έχει σχέση με τον πατέρα του και μέσω, μέσων που θα του επιτρέψουν ήδη από τους πρώτους μήνες της ζωής να βρίσκεται δίπλα στο παιδί που μόλις γεννήθηκε. Πιστεύω ότι πρέπει να απαντήσουμε και στις απαιτήσει της γυναίκας βεβαίω και στις απαιτήσει του πατέρα, αλλά να συνδέσουμε τις απαιτήσει αυτές με τις ανάγκες του νεογέννητου. Το παιδί χρειάζεται τον μπαμπά του. Γι' αυτό πιστεύω ότι η άδεια πατρότητας πρέπει να περιλαμβάνεται στο κείμενο αυτό και να είναι ένα στοιχείο θετικό αν λάβουμε υπόψη την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ γονέων και παιδιού. Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κανεί το λόγο. Θέλει το λόγο ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή. Κύριε Σότ. Όχι. ο κ. Λούντβικσον. Ούτε Σουηδέζα να ήσασταν. Λέω, ούτε Σουηδέζα να ήσασταν. Ευχαριστώ όσους συνέβαλαν στη συζήτηση για τις απόψεις και τις τοπολογίες που υπέβαλαν. Νομίζω οι περισσότερες είναι αποδεκτές, θα τις αναφέρω στην εισηγήτρια και ελπίζω να ξανακάνουμε και άλλη μια συζήτηση και να έχουμε όσο περισσότερες κοινέ συζητήσει εδώ. Υπάρχουν πολλές απόψεις εδώ, ελπίζω να βρεθεί λύση και βεβαίως εξαρτάται από όλους. Όταν μιλάμε για τις άδειε και το όλο των γυναικών στον χώρο εργασία, μιλάμε για πολύ σημαντικά ζητήματα αν τα δούμε, αν δούμε το μέλλον, αυτές, αυτά τα ζητήματα θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Και είναι σημαντικό να μπορέσουν να μετάσχουν στην αγορά εργασία οι γυναίκε αυτέ. Να ζητήσω συγγνώμη τώρα εξ ονόματο τη γειτονιά που δεν είναι εδώ. Έπρεπε να φύγει για να επιστρέψει στην πατρίδα τη για λόγου ενωτέρα βία. Θα τις περάσω πάντω ε, τι απόψει των συναδέλφων, ελπίζω να υπάρξει απόφαση πριν τον Ιανουάριο. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε βάση, κοινή βάση. Ευχαριστώ κύριε εισηγητή της εισηγήτριας. Είναι προφανές ότι υπάρχουν ε, αποκλίνουσες απόψεις ε, στο διάλογο, αλλά παρά τα αυτά πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να γίνει ο διάλογος αυτό σήμερα. Γιατί η επόμενη ενταλλαγή απόψεων θα έχει γίνει όταν ε, μετά από τις διμερείς και πολυμερείς συζητήσεις. Άλλωστε το Στρασβούργο είναι πάντα χρήσιμο γι' αυτό. 26 Ιανουαρίου θα τα πούμε. παρούσης της ηγήτριας και πρέπει να ψηφίσουμε και την επαύριο. Τελειώσαμε και αυτό το σημείο. Προτείνω να πάμε στο σημείο 6. Οργάνωση της ακρόασης που είχαμε ζητήσει να γίνει για την έκθεση Bauer σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών. Πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για να ξεκινήσει την ακρόαση αυτή, να υπενθυμίσω ότι Τώρα μπορούμε να έχουμε λίγη σιγή εδώ μέσα. Ζητήσαμε την άποψη της νομικής υπηρεσίας για τις συνθήκες εφαρμογής των υφιστάμενων δικαιωμάτων και χτες λάβαμε τη σχετική γνωμοδότηση. Η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου επιβεβαιώνει ότι οι, εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι εντάσσονται αυτόματα ή πάγονται αυτόματα στον, στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία 2015 ΕΟΚ από τι 20 Μαρτίου του 2009 και μετά. Λέω ξανά, Όσοι κουβεντιάζετε, να σηκωθείτε να φύγετε από την αίθουσα. Μα είναι φοβερό αυτό το φασαρία, μπουρου μπουρου μπουρου συνέχεια. Έλεγα λοιπόν ότι η νομική υπηρεσία υπογραμμίζει την ε, ρητή βούληση του νομοθέτη όπως εκφράστηκε από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου δηλαδή αυτού που αφορά το πεδίο επιφαρμογής, για την συμπερίληψη αυτή. Άρα η νομική υπηρεσία, επίση η νομική υπηρεσία υπενθυμίζει ότι οι ανεξάρτητοι οδηγοί, όπω ορίζονται στο άρθρο 3.1 σιγμα τη αυτής οδηγίας 2002-15 ΟΚ, υπάγονται αυτόματα στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγίας, ε, της οδηγίας και από τις 23 Μαρτίου του 9 οι υπόκεινται στις ρυθμίσεις του κειμένου αυτού ενώσο δεν τροποποιείται επί του σημείου αυτού ή εν λόγω οδηγία. Η νομική υπηρεσία αναφέρει επίσης ότι η έκφραση παρούσα οδηγία εφαρμόζεται δεν εκδηλώνει προγραμματική πρόθεση αλλά έχει επιτακτικό και άνευ όρων χαρακτήρα. Ιστορικά, η νομική υπηρεσία μας υπενθυμίζει ότι η νομολογία του ΔΕΚ για την εν λόγω οδηγία 2.15 ΕΟΚ. Έλεγα λέω στην οδηγία αυτή, είναι σαφές ότι η προσφυγή της, Ισπανία της Ισπανίας και της Φιλανδίας δεν θα ήταν παραδεκτή αν η συμπερίληψη των εξαρτήτων εργαζομένων στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία είχε ε, πραγματοποιηθεί υπό τον όρο τη πιθανή τροποποίησή τη. Τέλο, δύο κράτη-μέλη, Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία ήδη προέβλεψαν στην εθνική τους νομοθεσία την ε, εφαρμογή στους ανεξάρτητους από τις 23 Μαρτίου του 2009 Πρόκειται για ένα σημαντικό κείμενο που διαφωτίζει τις ανταλλαγές που θα κάνουμε, τις ανταλλαγές απόψεων που θα κάνουμε τώρα. Πριν δώσω το λόγο στους ε, προσκεκλημένους που καλωσορίζω, να σας πω ότι η ακρόαση γίνεται σε δύο τμήματα. Πρώτον, η κοινωνική εταίρη στενή ενία. Δεύτερον, τα ζητήματα ασφάλειας και επιμελητίας. Πριν, πριν θα δώσω όμως το λόγο στην κυρία Μπάουερ για να μας πει πώς θέλει να γίνει η συζήτηση. Έχετε το λόγο κυρία Συγκητρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητούμε το θέμα αυτό. Είναι προφανές ότι ακόμη τέσσερα σημεία συζητούνται και σε σχέση με τα τρία μπορούμε να βρούμε μια λύση. Για το τέταρτο όμως ακόμα συζητάτε. Είναι πολύ ευαίσθητο και το Κοινοβούλιο είναι χωρισμένο ως προς αυτό. Το πρώτο σημείο είναι η νυχτερινή εργασία. Νομίζω ότι αυτό θα, εδώ θα πρέπει να είμαστε πιο σαφείς. Να βρούμε έναν τρόπο να, είναι, να καταστεί το κείμενο πιο συγκεκριμένο για το χρόνο δηλαδή ο οποίος ουσιαστικά σημαίνει νυχτερινή εργασία. Πόσες ώρες είναι αυτή η νυχτερινή εργασία. και ελάχιστο να είναι το. Κάποιε απόψει λένε ότι ακόμη και ελάχιστο να είναι το διάστημα που δουλεύει κανεί το βράδυ, εξακολουθεί να θεωρείται νεκτερινή εργασία. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να είναι πολλέ οι ώρε. Ε, οι ώρες τώρα, αυτό, η πρόταση τώρα είναι για δύο ώρες. Πρέπει να βρούμε μια λύση ως προς αυτό. Ένα άλλο θέμα, ε, για το οποίο ακόμη δεν έχουμε βρει μια συμβαστική λύση, είναι το θέμα της εφαρμογής έχουμε κάποιες αμφιβολίες εδώ για το πού μπορούμε να, πού μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία. Ειδικά αν σκεφτούμε και το ωράριο εργασίας που μπορεί να μοιραστεί ανάλογα. Αυτό όντω πρέπει να το δούμε σε εθνικό επίπεδο, κατά πάσα πιθανότητα, σε επίπεδο δηλαδή εθνικής νομοθεσίας. Εκεί πρέπει να αναφέρονται όλα αυτά, να υπάρχει μια εσωτερική ρύθμιση. Πέρα από αυτό, στην οδηγία είναι σαφές ότι είναι απαραίτητο να φροντίσουμε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των αρχών για την επιβολή του νόμου. Ε, ένα άλλο καρφωτός θέμα είναι το τρίτο. Η, η ονή, ας πούμε, αυτοαπασχολούμενη. Εδώ θέλουμε ένα πιο συγκεκριμένο ορισμό των αυτοαπασχολούμενων η λέξη false είναι, έχει ε, αφαιρεθεί από το κείμενο. Η εμπειρία όμως δείχνει ότι εάν η οδηγία εφαρμοστεί από συγκεκριμένο κράτος μέλος, για παράδειγμα, στην Ουγγαρία, εμείς προσπαθούμε να εναρμονίσουμε τους κανονισμούς, τις οδηγίες. Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα σε αυτή την προσπάθεια όταν έπρεπε να ασχοληθούμε με τις πρωτοβουλίες κάποιων μεταρρυθμιστών υπουργών οι οποίοι πιέζουν ας πούμε για τις, ε, για τις νοσοκόμες ε, που, που θέλουν να θεωρούνται αυτοαπασχολούμενες σε κλινικές και νοσοκομεία. Βεβαίω αυτό ε, δεν μπορεί να δεν μπορεί να ισχύει ε, γιατί για παράδειγμα οι οδηγοί ε, φορτηγών αυτοκινήτων ε, μπορεί ας πούμε να πιεστούν και να αναγκαστούν να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι. Εγώ εκπροσωπώ αυτούς που λένε ότι θα πρέπει να στραφούμε στην Κομισιόν και να ζητήσουμε μια γενική έρευνα, μια μελέτη που θα αξιολογήσει την κατάσταση στην αγορά εργασίας γενικώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας ελέγξουμε ποιες οδηγίες και ποιοι κανονισμοί είναι ενισχύοι και ποιοι είναι εφαρμοστέοι. Διακόπτη η Πρόεδρος. Ε, ωραία, να το θέσουμε ως ερώτημα λοιπόν στους καλεσμένους μας. Ναι, σε σχέση και με την έκθεση αυτή, εγώ έχω πολλά θετικά παραδείγματα και θα ήθελα να ζητήσω από τους εμπειρογνώμονες ε, και τους ε, καλούς συναδέλφους να μου πούνε πώς ε, βλέπουν το θέμα αυτό των ιονί αυτοπασχολούμενων. Γιατί το θέμα τώρα είναι τι θα κάνουμε με τους αυτοαπασχολούμενους και τους ιονί αυτοαπασχολούμενους οδηγούς στην αγορά εργασίας. Γιατί αν εξαιρεθούν του πεδίου εφαρμογή και αν αυτή η έκθεση απορριφθεί, αν η οδηγία εξακολουθήσει να ισχύει, θα ξεκινήσουν 25 διαδικασίες επί παραβάση. Οπότε πραγματικά θα είναι σημαντικό πρόβλημα αυτό. Οπότε ας ρωτήσουμε τους ειδικού και επίσης θα ήθελα να μου πούνε τα αρνητικά και τα θετικά της εφαρμογής ή μη εφαρμογής της διάταξης αυτής στους ε, αυτοαπασχολούμενους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε τα ερωτήματα της εισηγήτριας. Σας προτείνω λοιπόν ακολουθήσετε αυτή τη γραμμή. Δηλαδή, πρώτα θα ακούσουμε τον κύριο Ρομπέρτο Παρίγιο, πρόεδρο του Τμήματος Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στις Μεταφορές και τον κύριο Μάρκο Ντίτζιο, Γενικό Γραμματέα Αναπληρωτή των ε, Οδικών Μεταφορέων Ξέρω ότι ήταν δύσκολο να βρεθεί, βρεθούν οι συνομιλητές, αλλά θα έχουμε δύο συνομιλητές σε αυτό το σημείο της συζήτησης. Δέκα λεπτά ο καθένας σας έχετε και στη συνέχεια θα ανοίξουμε τη συζήτηση με τους κοινοβουλευτικούς και θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι δεν έχετε αντίρρηση να ξεκινήσουμε με τον κύριο Παρίγιο. Πρόεδρο του Τμήματο Μεταφορών Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζόμενων στι Μεταφορές. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτέ, σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να τοποθετηθούμε. Θα κάνω μία σύνοψη του εγγράφου που είναι στη διάθεση όλων σας μετά την παρέμβασή μου. Λοιπόν, πριν από 7 χρόνια η οδηγία 2015 εγκρίθηκε για να ρυθμίσει το χρόνο εργασίας των εργαζόμενων στις οδικές μεταφορές. Τότε ο νομοθέτης πίστευε ότι ο προσδιορισμός των ελάχιστων προϋποθέσεων και χρόνου εργασίας ήταν απαραίτητος για να βελτιωθεί η ασφάλεια και η κατάσταση υγείας όσων ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα και επίσης για να υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός. Άλλαξαν τώρα οι περιστάσεις μετά από 7 χρόνια. Η σημερινή πρόταση υπονομεύει την ασφάλεια στους οδικούς άξονες. Ο κανονισμός 561 δεν αρκεί για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας. Η οδήγηση είναι η βασική δουλειά των οδηγών. Η πρόεδρος μιλάει χωρί μικρόφωνο δυστυχώ. Αν έχετε καλοσύνη, μην διαβάζετε πάρα πολύ γρήγορα. Ε, προσπαθείτε να κερδίσετε χρόνο, αλλά οι διερμηνεί ίσως δεν μπορούν να σα παρακολουθήσουν 100%. <laughs> Λοιπόν, εφόσον διαβάζετε πιο σιγά. Η Κομισιόν λοιπόν πιστεύει ότι η οδήγηση είναι η βασική απασχόληση των οδηγών. Συνεπώς αυτή η δραστηριότητα ρυθμίζεται από τον κανονισμό που αφορά την οδήγηση, το χρόνο οδήγησης και τον χρόνο ανάπαυσης. Πράγματι η οδήγηση μπορεί να είναι η βασική απασχόληση των οδηγών που καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις. Όμως αυτό δεν συμβαίνει για την διανομή, την παράδοση εμπορευμάτων, τις μεταφορές. Σε αυτή την περίπτωση η φόρτωση και η εκφόρτωση, ο χρόνος με τον πελάτη καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εργασίας του οδηγού. Σύμφωνα με την σημερινή πρόταση της Κομισιόν, οι οδηγοί, οι επαγγελματίες, οι ανεξάρτητοι έχουν στη διάθεσή τους 15 ώρες την ημέρα για να καλύψουν όλες αυτές τις δραστηριότητες και δεν πρέπει να τηρούν τον μέγιστο, το μέγιστο όριο οδήγησης. Και οι ανεξάρτητοι οι οποίοι οδηγούν οχήματα κάτω των 3,5 τόνων δεν έχουν ελάχιστο, μέγιστο όριο οδήγησης και ανάπαυσης διότι οι κανόνες δεν εφαρμόζονται σε οχήματα κάτω των 3,5 τόνων. Λοιπόν, ειδικότερα, σήμερα η μισθωτή οδηγεί μπορούν να εργαστούν, να φορτώσουν, να ξεφορτώσουν και να οδηγήσουν δηλαδή 48 ώρες την εβδομάδα ή μέγιστο 60 ώρες εάν σε μία περίοδο 4 μηνών ο μέσος όρος δεν ξεπερνάει 48 ώρες την εβδομάδα. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ένας μισθωτός που οδηγεί σήμερα 56 ώρες μια εβδομάδα μπορεί να αφιερώσει τέσσερις ώρες σε άλλες δραστηριότητες. Εάν το μεταφέρουμε αυτό στον ανεξάρτητο οδηγό μπορεί να οδηγήσει 56 ώρες και να έχει 30 ώρες άλλες δραστηριότητες σύμφωνα με την σημερινή πρόταση. Εάν υιοθετηθεί η πρόταση της Κομισιόν, ένας ανεξάρτητος οδηγός, ο οποίος παραδίδει εμπορεύματα σε διάφορα σούπερ μάρκετ παραδείγματος χάρη, και είναι μία περίπτωση σύνηθης για μέσες ε, αποστάσεις, κάθε μέρα έχει 13 με 15 ώρες για να φορτώσει και να εκφορτώσει, για να οδηγήσει το φορτηγό του και τι ασφάλεια υπάρχει συνεπώς για τους πολίτες που πηγαίνοντας στη δουλειά τους ή στο σχολείο ή διασχίζοντας το δρόμο θα μοιράζονται τους δρόμους με οδηγούς φορτηγών που εντός εισαγωγικών θα, θα εργάζονται 13 με 15 ώρες την ημέρα ή αν όχι παραπάνω. Γι' αυτό η Ομοσπονδία μας θεωρεί ότι η σημερινή πρόταση της Κομισιόν δεν εξασφαλίζει την ασφάλεια στους αυτοκινητοδρόμους και στους δρόμους της Ευρώπης. Η σημερινή πρόταση υπονομεύει τον θεμητό ανταγωνισμό θα αποτελέσει κίνητρο για τις οδικές μεταφορές να, μετατραπού να μετατρέψουν τους επαγγελματίες οδηγούς τους σε αυτοαποσχολούμενους. Έχουμε πολλαπλασιασμό λοιπόν αυτών των περιστατικών, αλλά προς το παρόν υπάρχει ένας περιορισμός χάρη στην κλαδική οδηγία. Η οδηγία 2002 κάθετος 15 ε, προσδιορίζει τις προϋποθέσεις για τους αυτοαποσχολήμονους ε, οδηγούς. Τώρα, όσον αφορά τις τις επιδράσεις, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ανάμεσα στα πιο συχνά επιχειρήματα για να αντιταχθεί κανείς στη ρύθμιση του χρόνου εργασίας είναι εκείνο που λέει ότι η συμπερίληψη των ανεξαρτήτων ε, οδηγών θα επηρεάσει καταστροφικά τις μικρομεσαίες που είναι η μεγάλη πλειοψηφία των μεταφορικών εταιριών όταν έχουν ένα-δύο οδηγού δεν επηρεάζονται διότι είναι μισθωτοί οι οδηγοί. Άλλα συμφέροντα κινδυνεύουν οι μικρομεσαίε επιχειρήσεις οδικών μεταφορών είναι τόσο ζωτικές ε, και τόσο πολύ άριθμες, όχι επειδή έχουν μεγάλα κέρδη μέσα στο διαρκές επιχειρηματικό πλαίσιο, αλλά διότι προσφέρουν χαμηλό κόστος υπηρεσίας και οι πρακτικές τους είναι πολύ πιο δύσκολο να ελεγχθούν. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η μεγάλη πολυεθνική Ρενό έχει υπεργολάβους μικρούς οι οποίοι εφαρμόζουν συνθήκες dumping. Είχαμε πολλά τέτοια παραδείγματα αυτή την εβδομάδα. Η DHL, η DHL είναι άλλη τέτοια περίπτωση. Οι μικρομεσαίες που θα χρησιμοποιούσαν τους ε, ανεξάρτητους οδηγούς μπορεί βεβαίως να κάνουν μια οικονομία. Αλλά η πρόταση σημερινή δεν είναι αποτελεσματική διότι ως προς τον, θε, τον θέμητο ανταγωνισμό παραγνωρίζει τις συνθήκες βάσει των οποίων οι αυτοαποσχολούμενοι μπορεί να δηλώνονται σε μια χώρα αλλά να, χώρα, να εργάζονται σε άλλη. Οπότε ο έλεγχος αυτών των αυτοαποσχολούμενων ε, δεν θα είναι εφικτός παρά μόνο στη χώρα όπου έχουν δηλωθεί, ενώ αυτοί θα εργάζονται αλλού. Συνεπώς, η πρόταση της Κομισιόν δεν μας δίνει κανένα μηχανισμό ελέγχου που, ώστε να αποφύγουμε το κοινωνικό dumping στις οδικές ε, μεταφορές. Γι' αυτό παρατηρούμε ότι υπάρχουν μεγάλες αλήψεις στην πρόταση. Επίσης, επηρεάζει την ασφάλεια και την υγεία των επαγγελματιών οδηγών και επιβαρύνει και το κόστος. Γι' αυτό η Ομοσπονδία μας ελπίζει ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα υιοθετήσει τη δικιά μας λογική. Τι προτείνουμε. Θέλουμε μία κλαδική οδηγία για τη ρύθμιση του χρόνου εργασίας με πεδίο εφαρμογής όλους τους επαγγελματίες οδηγούς. Μία οδηγία η οποία να διευκρινίζει τα μέτρα ελέγχου για τους αυτοαπασχολούμενους και να υπάρχει και η αρχή συνυπευθυνότητας όπως το άρθρο 10 του 561. Έτσι θα εφαρμοστεί καλύτερα ο κανόνας του χρόνου εργασίας και η ευθύνη της μη τήρησης των διατάξεων του κανονισμού θα χρεώνεται και στον αυτοαποσχολούμενο αλλά και στον πελάτη και στον εργοδότη. Παραγγέλλοντα μάλλον. Πρέπει να δουν επίσης τις τάσεις στα κράτη-μέλη σε αυτό το κλάδο, να δουν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από τον αθέμητο ανταγωνισμό και επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια. Με αυτές τις εκθέσεις λοιπόν που θα λάβει η Κομισιόν από τα κράτη-μέλη μπορεί να κάνει μια σύνοψη προς το Συμβούλιο και να υπάρξει μια πραγματική διασύνδεση μεταξύ οδηγίας και του κανονισμού για το ταχύμετρο ώστε να μπορεί να παρακολουθηθεί ο χρόνος εργασίας. Έχουμε το σχετικό κανονισμό που θα αναθεωρηθεί το 2010. Θέλουμε λοιπόν μια οδηγία που να εφαρμόζει ένα αναγκαστικό σύστημα χρόνου εργασίας. Ας διευκρινίσουμε ακόμη ότι θα θέλαμε η διοικητική εργασία των αυτοαποσχολούμενων, η λογιστική και οι σχέσεις με τον ε, πελάτη να μην περιλαμβάνονται στο χρόνο εργασίας. Ο χρόνος εργασίας να συσχετίζεται μόνο με τη μεταφορά. Δεν θέλουμε να περιορίσουμε τον χρόνο εργασίας των ανεξαρτήτων, των αυτοαποσχολούμενων, αλλά να δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο, πλαίσιο το οποίο να τηρείται από κάθε επαγγελματία οδηγό. Πρώτη φάση αυτή. Θέλουμε όμως ένας νέος κανονισμός να ασχοληθεί και με τους ψεύτο ανεξάρτητους. Πολύ σημαντικό αυτό για μας, για να οριστεί ένα γενικότερο πλαίσιο. Καταλήγω λέγοντας ότι υπάρχουν τρία στοιχεία τα οποία πρέπει να συνδεθούν οπωσδήποτε. Η ασφάλεια, η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία και ο θεμητός ανταγωνισμός. Δεν θέλουμε να επιτεθούμε στους αυτοαπασχολούμενους. Αντίθετα, θέλουμε να να εξασφαλιστεί η ασφάλεια η οδική όλων των Ευρωπαίων, η υγεία και οι συνθήκες εργασίες για όλους τους οδηγούς και ο θεμητός ανταγωνισμός που είναι ο βασικός κανόνας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτά τα πολύ σημαντικά στοιχεία που μας δώσατε. Ο κύριος Μάρκο Τιγκιουίλα θα μας μιλήσει τώρα. Είσαστε Γενικός Γραμματέας της UTR και νομίζω ότι έχετε και ένα δεύτερο ε, καπέλο με τις μικρομεσαίες οδικών μεταφορών. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Μπάουερ για την πρόσκλησή της να συμμετάσχουμε. Η UTR ευχαρίστω συμβάλλει σε αυτή τη συζήτηση και θα ήθελα να σας δώσει τις απόψεις της σε σχέση με την επεξεργασία από την Επιτροπή σας της τροποποίησης της οδηγίας 2002 κάθετος 15. Εκπροσωπούμε περίπου 200.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον ε, τομέα των μεταφορών από την ανατολική και δυτική πλευρά και μετά από τις πρόσφατες συζητήσεις που γίνανε στο Ευρωκοινοβούλιο για την ε, οδηγία 15 ζητάμε λοιπόν τον αποκλεισμό των ε, αυτοαποσχολούμενων οδηγών και θα σας εξηγήσω γιατί. Πρώτα απ' όλα, οδική ασφάλεια. Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας είναι μεγάλο θέμα για τις μεταφορικές εταιρείες. Ο κύριος Παρίο πριν αναφέρθηκε στο πρόβλημα των μικροτέρων οχημάτων. Αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ένας νέος κανονισμός 68 του 2009 του Ιανουαρίου φέτος προσάρμοσε για ένα τη φορά τον κανονισμό του Συμβουλίου και τώρα περιλαμβάνει και τα μικρότερα οχήματα, την εγγραφή τους και τα λοιπά. Και υπάρχει συγκεκριμένο ταχυγράφος για αυτά τα οχήματα, δεν είναι ακριβώς ταχυγράφος, είναι ένα άλλο μηχάνημα καταγραφής. Όσον αφορά τα οδικά ατυχήματα, είναι ο τομέας μας, ο κλάδος μας είναι ασφαλέστατος στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τις τελευταίες στατιστικές του παρετηρίου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μόνο 2,8 κάτω από 3% ε, ατυχήματα με επαγγελματικά οχήματα κάτω των 3,5 τόνων που είναι ακριβώς αυτά που χρησιμοποιούν οι αυτοαποσχολούμενοι. Λοιπόν, κάτω από 3% σας παρακαλώ, σημειώστε, σημειώστε το ε, και όλα αυτά τα στοιχεία αφορούν το 2008. Τώρα, η υγεία των οδηγών είναι ένα άλλο θέμα που μας ενδιαφέρει. Αλλά επιτρέψτε μου και εδώ να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία. Όσον αφορά μια έκθεση του 2007 η υψηλότερη έκθεση σε μακρές ώρες εργασίας αναφέρονται στην αλληλεία και στη γεωργία και στις οικοδομές. 40% ήταν το ύψος. Ενώ ε, στις μεταφορές έχουμε κάτω από 5% τέτοιες περιπτώσεις. Δεύτερος τώρα λόγος πυροχηματολογίας. Ας θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο ε, για τη δραστηριότητα αυτών των αυτοαπασχολούμενων. Έχουν οικονομικό κίνδυνο. Λοιπόν, και θα τους αποκαλέσω τους αυτοαποσχολούμενους επιχειρηματίες τρόπον την άδεια, διότι έχουν να αντιμετωπίσουν οικονομικό επιχειρηματικό κίνδυνο. Λοιπόν, αν εφαρμοστεί η οδηγία έτσι όπως έχει σε αυτούς τους οδηγούς, θα περιοριστεί η εργασία τους. Ε, οι οδηγοί που είναι εκτός ΕΕ θα μπορούν να εργαστούν περισσότερες ώρες. Επίσης, οι διατάξεις αυτές θα υπονομεύσουν αυτούς τους οδηγούς τους αυτοαπασχολούμενους σε σχέση με άλλους αυτοαπασχολούμενους, σε άλλο κλάδο. Αυτό θα αποτελέσει πολύ επικίνδυνο προηγούμενο στον περιορισμό των δικαιωμάτων τους. Η UTR πάντα έλεγε ότι το πρόβλημα dumping αφορά βασικά το κόστος. Τα μεταφορικά είναι πολύ χαμηλότερα σήμερα από το πραγματικό κόστος της μεταφοράς. Δηλαδή δεν παρέχουν τη δυνατότητα για ένα ελάχιστο εισόδημα. Μιλώ πραγματικά για την επιβίωση αυτών των ανθρώπων. Όπως ξέρετε, ο μεταφορικός κλάδος είναι σε μεγάλη κρίση, όπως τόσοι άλλοι κλάδοι. Ε, πτώση της ζήτησης, κλείνουν οι πελάτες κτλ. Και όλα αυτά επηρεάζουν σημαντικά την πραγματική οικονομία. Έτσι πέφτει δεν εκδίδονται νέες άδειες, έχουμε μεγάλη πτώση και έχουμε και αύξηση στην ανεργία. Και το ΑΕΠ δεν προοδεύει. Υπάρχουν διαρθρωτικές αδυναμίες, καθυστέρηση στην εξόφληση δανείων, προθεσμίες ε, ε, 30 ημερών που δεν εφαρμόζονται πια, όλα αυτά αυξάνουν το κόστος και συνεπώς η οδηγία μαζί με όλα τα υπόλοιπα τελικά θα αφαιρούσε κάθε ίχνος οξυγόνο από αυτό το επάγγελμα. Ε, είναι μεγάλη υπόθεση βεβαίως για ε, αυτά αυτό απασχολούμενοι οδηγοί. Αυτό είναι αλήθες, ότι υπάρχουν ε, ψεύτο αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί για πολλούς λόγους. Αλλά αν πάρετε την εμπειρία πολλών κρατών μελών θα δείτε ότι στρατηγικές δεν επικεντρώνονται στο χρόνο εργασίας. Υπάρχουν νέοι μηχανισμοί που αναπτύσσονται για την αντιμετώπιση παρανόμων καταστάσεων με τη βοήθεια και των επαγγελματικών οργανώσεων. Τέλος, τελευταίο επιχείρημα, η παρακολούθηση, η εποπτεία. Οι αυτοαποσχολούμενοι είναι αδύνατο να διαχωρίσουν τον χρόνο εργασία τους από τον υπόλοιπο χρόνο. Ε, είναι λιγότερο δομημένος ο χρόνος εργασίας τους λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους. Επίσης είναι αδύνατο να παρακολουθήσουν και να καταγράψουν αυτόν τον χρόνο ή να το κάνει κάποιος άλλος. Η οδηγία προβλέπει υποχρεωτική καταγραφή των ε, ωρών, του χρόνου μάλλον. Επίσης, αυτός ο αυτοαποσχολούμενος δεν έχει τη διοικητική υποδομή για να τα κάνει όλα αυτά. Δηλαδή να έχει ε, οδηγεί, να έχει τι επαφέ με τον πελάτη ε, και να καταγράφει και να ε, κρατά όλα τα έγγραφα. Επίσης, η δίωξη θα είναι αδύνατη. Οι δημόσιες αρχές που πρέπει να φροντίσουν για την εφαρμογή δεν έχουν ιδέα πώς να προχωρήσουν στην εφαρμογή μιας τέτοιας οδηγίας είναι ανέφικτο δηλαδή. Καταλήγοντας, η UTR θέλει μια ρεαλιστική και συγκεκριμένη προσέγγιση. Θέλει την υγεία, την οδική ασφάλεια και την ευρωπαϊκή ένταξη. Όμως, η εμπειρία στον τομέα και η σημερινή οικονομική κρίση πρέπει να ληφθούν υπόψη από το Ευρωκοινοβούλιο. Μια υγιής ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να είναι αποτελεσματική υποστηρίζοντας το ρόλο αυτών των αυτοαποσχολούμενων οδηγών. Να ενισχύσει τον ανταγωνισμό και να μειώσει τις διοικητικές επιβαρύνσεις. Έχουμε ολόκληρη κρίση να αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους δύο προσκεκλημένους μας. υπήρξε κάποιο πρόβλημα εκπροσώπησης ορισμένων ε, που είναι δευτερότερο έχω τρεις ε, που έχουν ζητήσει τρεις ε, που έχουν ζητήσει το λόγο δεν έχουμε πολύ χρόνο να τσεκάρω ποιοι θέλουν να μιλήσουν τέσσερις δεν, χρειάζεται να μιλήσετε και καλά όλοι, γιατί είσαστε, όσο περισσότεροι είσαστε, τόσο λιγότερο χρόνο έχει ο καθένα στη διάθεσή του. Ωραία. 1,5 λεπτό ο καθένα. Ο κύριο Φάμπρο και μετά ο κύριο Κοφεράτη. Κύριε Φάμπρο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Να σας πω εισαγωγικά ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπαν οι εκπρόσωποι των συνδικάτων. Γιατί δημιουργήθηκαν οι, ανεξά, οι, οι εργαζόμενοι. Γιατί οι εργοδότες δεν θέλουν να πληρώνουν την συνεισφορά τους ούτε την ασφάλεια, ε, την ιατρική ασφάλεια. Εγώ δεν συμφωνώ με το ότι κάποιος πρέπει να δουλεύει όσο θέλει. Είναι παράλογο. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι νόμοι που θα προστατεύουν τον άνθρωπο από τον εαυτό του. Όλοι ξέρουμε ότι το, το ξέρουμε αυτό. Ήδη το 1919 εγκρίθηκε η πρώτη σύμβαση για τη μέγιστη διάρκεια εργασίας. Δεν συμφωνώ ότι όσοι δουλεύουν επιμακρό δεν θέτουν σε κίνδυνο τους συμπολίτες στο δρόμο. Τα ατυχήματα που γίνονται στη χώρα μου, την Τσεχία, το επιβεβαιώνουν αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εξαιρετικά κουρασμένοι και δεν μπορούν να κρατήσουν στο δρόμο. Δεν είναι δυνατόν. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να δεσμεύσουμε, να του βάλουμε κάποιου να δουλεύουν σαν σκλάβοι συνέχεια. Ο κύριος Κοφεράτη. Ευχαριστώ. Εγώ πιστεύω ότι η ασφάλεια είναι ένα σύγχρονο δικαίωμα ηθαγένειας που πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους ανθρώπους όσο καλύτερα γίνεται. Επίσης, πιστεύω ότι αποτελεί μια προτεραιότητα με την οποία να συνδέσουμε τις βράσεις που πρέπει να αναλάβουμε. Προσπαθώντας, δεν μπορούμε να, λύσουμε τα προβλήματα, δεν κάνουμε μια αντιπαράθεση ένα κλάδο. Διότι όπου υπάρχει κίνδυνος υπάρχει πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε. Όταν μιλούμε λοιπόν για ωράριο δεν μπορούμε παρά να ξεκινήσουμε από αυτή τη βάση. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι θεμελιώδες να επεκταθεί ο ίδιος κανόνας σε όσους εμπλέκονται στην δραστηριότητα αυτή. Είτε είναι υπάλληλοι, είτε είναι ανεξάρτητοι. Δεν ξεχνάω το πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή της δουλειά των ανεξαρτήτων. Αλλά τα προβλήματά τους κάτω από μια κατάσταση κρίσης πρέπει να αντιμετωπιστούν με ενισχύσεις, με συγκεκριμένες ε, δράσεις, αλλά ποτέ δεν πρέπει να συνδέονται με μορφές που θέτουν σε κίνδυνα την ασφάλεια. Να προσθέσω ότι αν δεν υπάρξει ομοιόμορφη αντιμετώπιση, μπαίνουν ε, αλλαγές στη δυναμική του ανταγωνισμού και εν τέλει αυτός που συμπεριφέρεται άσχημα πληρώνει λιγότερο από ό,τι από αυτός που πληρώνει, που τηρεί τους κανόνες. Η κυρία Τούρινεν πρώτα. Ευχαριστώ. η συζήτηση έχει διαιρεθεί. Θα ήθελα να ζητήσω από τους εκπροσώπους των συνδικάτων να μας πούν τι είχαν, γιατί εγώ τις διάβασα πριν έρθω, αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί θα μου πάει πάρα πολύ χρόνο. Θέλω να, ρωτήσω μία, να θέσω μία ερώτηση για, τα θέμα, για το ζήτημα των ελέγχων. Πολλοί λένε ότι Εάν συμπεριλάβουμε στον εγκανονισμό και τους αυτοπασχολούμενους δεν θα μπορέσουμε να το ελέγξουμε. Αυτό ωστόσο δεν ισχύει. Και ο κύριος Κράμες δική του παρουσίαση που θα την ακούσουμε σε λίγο έγραψε ότι ναι μεν αυτοί δεν κρατούν ώρες εργασίας αλλά τις κρατάει που ισχύει και για τις δύο κατηγορίες. Ο ψηφιακός ταχογράφος αρχίζει να δουλεύει με το που ανοίγει τη μηχανή είτε είναι ε, ε, μισθωτός είτε είναι ανεξάρτητος εργαζόμενος. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν υπάρχει δυνατότητα εφόσον μπορούμε να ελέγξουμε με τον ταχογράφο αυτό το σύστημα ε, γιατί λέτε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους ανεξάρτητους. Μετά το άλλο ζήτημα είναι η εικονική αυτοαπασχολούμενη. Πώς ορίζεται αυτό νομικά. να τελειώ, θέλω να τελειώσω πρώτα, το ξέρω. Δηλαδή μιλώ για ανθρώπους που ναι φαίνονται αυτοαπασχολούμενοι αλλά είναι υπάλληλοι στην πραγματικότητα. Μήπως δημιουργήσουμε μια τρίτη κατηγορία ε, εργαζομένων. Κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε πάρα πολύ σύντομα. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να επεκταθεί η νομοθεσία και στους αυτοαποσχολούμενους. Δεν είναι μόνο ένα θέμα εργασιακό και ωραρίου. Είναι θέμα που αφορά την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Ξέρουμε ότι οι οδηγοί αυτοί ουσιαστικά έχουν άμεση σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όταν από τη μια μεριά θέλουμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από την άλλη επιθυμούμε να έχουμε, να δώσουμε ένα κοινωνικό πρόσωπο στην Ευρώπη, Όλα αυτά πρέπει να τα συνδυάσουμε μέσα στο πλαίσιο της νομοθεσίας. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι δίνουμε ένα κοινωνικό παράδειγμα εάν προωθήσουμε την ένταξη και των αυτοαπασχολουμένων. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρονή μετά Χάντερ. Ευχαριστώ για την ασφάλεια και υγιεινή στον χώρο εργασία των εργαζόμενων σε οδικέ μεταφορέ δεν θα επανέλθω γιατί συμφωνώ με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι προηγουμένω. Στη Γαλλία διαπιστώνουμε ότι η μείωση του χρόνου εργασία στου οδηγού μείωσε κατά πολύ τον αριθμό των ατυχημάτων. Σε ό,τι αφορά του ανεξάρτητου, ιδίω δε του πλασματικού ανεξάρτητου, ε, υπάρχει μια σοβαρή διαπίστωση αθέμητου ανταγωνισμού από χώρα σε χώρα μεταξύ χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν πρέπει να του αποκλείσουμε. Σε ό,τι αφορά του ελέγχου, δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη παρά μόνο το χρόνο οδήγηση και των συναφών ε, δραστηριοτήτων και όχι όλε τι δραστηριότητε. Οι ταχογράφοι μπορούν να λάβουν υπόψη το ακριβώ αυτή την διάσταση και την περίοδο. Δεν υπάρχει κανένα μέσο που να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον διαπιστώνω ότι πολλέ επιχειρήσει στη Γαλλία δημιουργούν πλασματικού ανεξάρτητου σε άλλα κράτη-μέλη. Κάτι που θα πρέπει οπωσδήποτε να λύσουμε. Αυτά και περιμένω, ελπίζω από τους συναδέλφους να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό. Ευχαριστώ. Πολλά σχόλια, πολλές ερωτήσεις για τους ε, ε, προσκεκλημένους μας. Ο κύριος Τόμας Χέντελ είναι τελευταίος ερωτών. Ένα ερώτημα, Πρόεδρε. Ρωτώ και τους δύο εμπειρογνώμονες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 ένα α πούμε Ισπανός οδηγό θέλει να ε, ελέγξει έναν Ρουμάνο και βλέπει ότι ε, έχουν ε, τηρηθεί οι ώρε εργασία χωρί να υπάρχει νομική βάση για το αν είναι αυτοαπασχολούμενο ή υπάλληλο. Πώ μπορούν να μου απαντήσουν οι πυρογνώμονε. Δεύτερον, ελπίζω να συμφωνούν οι πυρογνώμονε μαζί μου ότι το ωράριο και η πολιτική για το ωράριο είναι πάντα πολιτική, κοινωνική και ήταν πάντα κομμάτι της κοινωνική πολιτική. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι περίπου περίεργο να λέμε τώρα υπάρχει διακριτική μεταχείριση των αυτοποσχολούμενων αν μπουν σε μια νομική διάταξη ε, που περιλαμβάνει και πτυχές ε, υγείας και ασφάλειας. με, σύμφωνα με την άποψη της Κομισιόν δηλαδή πρέπει να έχουμε 68 α, ώρες οδήγησης και ε, φορτοεκφόρτωσης και μετά άλλες 20 ώρες έξτρα τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, και αυτό τι είναι, είναι ανθρώπινο αυτό το ωράριο δηλαδή, εσείς πώς το βλέπετε. Τρίτον, αυτό που είπε ο κύριος Κονφεράτη θα υπάρξει μεγάλη στρέβλωση του ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά του αυτοαποσχολούμενου με αυτέ τι ώρε οδήγηση, σε ό,τι αφορά το, το, dumping μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων, γιατί θα είναι τελείω διαφορετική η κατάσταση με του υπαλλήλου. Αυτό θέλετε να κάνετε στο μέλλον ή θέλετε να υποστηρίξουμε αυτό μέσω της πρόταση Κομισιόν. Ευχαριστώ. Θα δώσω δύο λεπτά στους προσκεκλημένους μας, δύο λεπτά στον καθένα από τους προσκεκλημένους μας για να απαντήσουν. Διτζόη, ο κύριο Διτζόη πρώτο. Ε, merci beaucoup. Ε, allow me to θα απαντήσω στη μητρική μου γλώσσα, τεταλικά. Ε, Σε ό,τι αφορά τα τελευταία τρία ερωτήματα που μου απευθύνθηκαν. Ένα. Για τον έλεγχο στη Ρουμανία, για παράδειγμα τις εργασίες ε, ενός μιας ισπανικής επιχείρησης μπαίνει στο παιχνίδι και μια άλλη βασική διάσταση του θέματος. Κατάρτιση και εφαρμογή ελέγχων. Σε πολλά κράτη-μέλη οι εθνικές ε, οργανώσεις μεταφορών είναι οι πρώτες που ζητούν αύξηση των ε, ελέγχων και χρηματοδότηση των ελέγχων από πλευρά εθνικών αστυνομικών αρχών επί των ίδιων των επιχειρήσεων. Σας διαβεβαιώνω ότι είναι πολύ δύσκολο γιατί τα κράτη-μέλη και οι κυβερνήσει δεν θέλουν να χρηματοδοτούν και να κατατρίζουν τις αστυνομικέ του δυνάμει. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το ωράριο εργασία και το συσχετισμό του ωραρίου με την υγεία αναφέρθηκα πριν από λίγο σε στατιστικές ε, τελείως αμερόληπτες που υπογραμμίζουν ότι είναι άλλοι οι τομείς όπου ο κίνδυνος υγείας από την υπερβολική δουλειά είναι παρόν. Τέλος, σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα, επαναλαμβάνω εκ νεού ότι το πραγματικό πρόβλημα του κοινωνικού ντάμπινγκ αφορά τις επιχειρήσεις μεταφορών που προσλαμβάνουν οδηγούς που πληρώνονται πολύ λιγότερο από τις αμοιβέ που, που δίδονται σε άλλα κράτη-μέλη και που ζουν κάτω από συνθήκες εργασίας οι οδηγοί φρικτές. Διότι αν δεν υπάρχουν ε, πάυσεις ε, οδήγησης και αν υποχρεώσω τον, ε, τον οδηγό να μεταφέρει το εμπόρευμα σε απίθανες ώρες εκτός αν τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα δημιουργώ βλάβη και στην ζημιά και στην οδική ασφάλεια. Άρα υπάρχει ταυτόχρονα και κοινωνικό ντάμπινγκ και αύξηση της οδικής ανασφάλειας. Συγγνώμη που σας βάζω σε αυτό τον φρικτό ρυθμό απάντησης που είναι το Κοινοβούλιο. Δύο λεπτά. Και εσείς κύριε Παρίλο. Επί του ελέγχου. Υπάρχει μία πρόταση ρεαλιστικής συζήτησης που αφορά τον έλεγχο και των δύο καθεστώτων. Πρώτον, ο... για... πρέπει να υπάρχει έλεγχος συνυπεύθυνος για να ελέγξουμε του, τους πρέπει να πάμε στην επιχείρηση. Για να ελέγξουμε τους ανεξάρτητους πρέπει να ελέγξουμε τον ίδιο τον ανεξάρτητο. Τον, να πάμε στο αυτοκίνητο. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα ατύχημα πρέπει να βρούμε κατά πόσο ο οδηγός είναι υπεύθυνο ή όχι. Και μετά μπαίνουμε, έτσι μπαίνουμε στην ευρωπαϊκή οπτική μείωση του, του διοικητικού βάρους. Δεύτερον, νομικά. Τι μας λένε όταν έχουμε έναν πολίτη είμαστε πλασματικοί ανεξάρτητοι. Θα δαπανίσουμε χρήματα στην Ευρώπη για να πάμε να δούμε πόσους πελάτες έχουμε με το Υπουργείο Οικονομίας, με, το Ομοσπονδιακό, ε, με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μεταφορών, το Υπουργείο Μεταφορών και ε, βρίσκουμε έναν πελάτη, του λέμε είσαι ψευτο ανεξάρτητος, αλλά όταν έχεις δέκα πελάτες είσαι πραγματικό ανεξάρτητο. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Πρέπει να λάβουμε λοιπόν υπόψη αυτό, πρέπει να λάβουμε υπόψη την υγιεινή και την ασφάλεια, αλλά και τα ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό dumping. Σήμερα στην Ευρώπη, όταν ένα Γάλλος οδηγό κερδίζει 100 ευρώ, ο οδηγό ο Ούγκρος παίρνει 36. Και αν φροντίσουμε να και ότι και αν ε, πάμε με πλασματικού ανεξάρτητου από τη μια χώρα στην άλλη, έλεγχο πραγματικό δεν γίνεται. Γιατί κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για του δικού τη ανεξάρτητου, όχι για του ανεξάρτητου άλλων χωρών. Άρα, με τι προτάσει αυτέ, δημιουργούμε την βάση μια, ενός αφέμητου ανταγωνισμού και τη διάλυση του τομέα των μεταφορών. Γι' αυτό λέμε πρώτη οδηγία που θα περιλαμβάνει όλους τους ανεξάρτητους οδηγούς και μετά ένας κανονισμός που θα αφορά πολύ κλαδικά τους πλασματικούς ανεξάρτητους. Αλλά ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη ανεξάρτητα, ενώ η οδηγία ενσωματώνεται στα κράτη-μέλη και ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τους πλασματικούς ανεξάρτητους. Εγώ θέλω να λάβουμε υπόψη όλους τους εργαζόμενους στον τομέα. Ευχαριστώ. Πάμε στο δεύτερο τμήμα της ακρόασης που αφορά περισσότερο ζητήματα επιμελητίας και ασφάλειας. Δίνω το λόγο στον κύριο Χένκε Κράμερ, υπεύθυνο ευρωπαϊκών υποθέσεων και για τις μεταφορές στην Ολλανδία. Δέκα λεπτό το maximum. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την ε, δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω για ένα θέμα που έχει τύχει πολλών συζητήσεων το τελευταίο χρόνο. Εγώ εργάζομαι στον τομέα αυτό από το 1979 και από τότε το κουβεντιάζουμε. Κάποια συμπεράσματα να σας αναφέρω. Εγώ εκπροσωπώ την TLN, το ε, Ολλανδικό Συνδικάτο για τους ε, Οδηγούς. Ε, εκπροσωπούμε περίπου 60.000 ε, επιχειρήσεις, πολλές μεγάλες, πάρα πολλές μικρές. Έχουμε 1.500 εταιρείες μεταφορών που είναι ανεξάρτητες και είναι πολύ περήφανες που είναι ανεξάρτητες και είναι μικρές, μικρού μεγέθους επιχειρήσεις. Θέλουν να παραμείνουν μικρές επιχειρήσεις. Βέβαια εντάξει κάποιες φορές εξαγοράζονται από μεγαλύτερες αλλά όλοι ξεκίνησαν με ένα φορτηγό κάποτε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Να σας αναφέρω κάποια στοιχεία σε σχέση και με την θέση του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Μεταφορών. Καταρχήν, το ωράριο για τους μετακινούμενους εργαζόμενους δίνει κοινωνική προστασία για τους εργαζόμενους και αυτό είναι πάρα πολύ καλό είναι μεγάλο επίτευγμα για όλους. Τώρα, η ETF ε, τώρα ε, υπερασπίζεται τα δικαιώματα των αυτοαπασχολούμενων. Ξαφνικά δηλαδή υπάρχει ανάγκη να αλλάξουν τα πράγματα. Γιατί? Γιατί ξαφνικά έχει γίνει τόσο μεγάλη αλλαγή. Ε, έχει υπάρξει μεγάλη αλλαγή και στον τομέα ε, που μας οδήγησε στο να κάνουμε και εμείς τέτοιου είδους αλλαγές και με το ε, προηγούμενο των, ε, της ασφάλειας των αυτοπασχολούμενων έναντι των υπαλλήλων, τι γίνεται, βελτιώθηκε ή χειροτέρευσε. Έχουμε κάποια στατιστικά στοιχεία εμείς, λίγα μεν, αλλά παρόλα αυτά, αυτά τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο. Οι οδικές μεταφορές έχουν γίνει πιο ασφαλείς χάρη στις ε, ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, σε εθνικές πρωτοβουλίες και σε τομεακές πρωτοβουλίες. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα, Έχουμε τον νέο βελτιωμένο κανονισμό για τις ώρες οδήγησης, τις ώρες ε, ε, ανάπαυσης, του ταχογράφου που θα είναι βελτιωμένοι και θα είναι διαθέσιμοι στους ε, επαγγελματίε του τομέα αυτού και αυτό βοηθά στο να αυξηθεί η οδική ασφάλεια. Οπότε η ETF λέει ότι οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί εργάζονται 84 με 86 εβδομάδα, ε, ώρες την εβδομάδα, ε, κάθε εβδομάδα το χρόνο. Γιατί ο 561 του 2006 για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης δεν είναι κοινωνικός κανονισμός. Οι παρενέργειες είναι ότι περιορίζει τις ώρες εργασίας, εργασίας και ώρες οδήγησης για τους ε, αυτοπασχολούμενους. Είναι αδύνατο λοιπόν να υπάρχει εβδομάδα με 84 ώρες ή 86 ώρες οδήγησης. Η ETF λοιπόν αξιολογεί την κατάσταση των ε, υπαλλήλων οδηγών, οι οποίοι μετά μετατρέπονται σε ε, πλασματικούς ε, αυτοπασχολούμενους. Πολλά έχουν αντιμετωπίσει επιτυχώς το θέμα αυτών των πλασματικών ή αυτοπασχολούμενων οδηγών. Και να πω και κάτι για τις αρχές για τις οποίες ε, συζητούμε. Υπό το φως τη της άποψης της TLN και άλλων οργανισμών στις ε, χώρες μέλη της Ένωσης, η συμπερίληψη των, ε, των αυτοαπασχολούμενων στον κανονισμό για τις ώρες εργασίας αντίκειται σε όλα όσα πρεσβεύουμε. Δηλαδή μπορείτε να ρυθμίσετε τις ώρες Εργασία ε, το ωράριο ενό καταστήματο. Εντάξει, αυτό μπορείτε να το κάνετε, ε, μπορείτε να το κάνετε και για τους ε, ηλεκτρολογού και για τους χειρουργού και για τους ανεξάρτητους οδηγού. Δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο νομοθεσίας για τους επιχειρηματίε. Και νομίζω ότι αν προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση θα, θα δημιουργήσουμε ένα κακό προηγούμενο. Η συμπερίληψη λοιπόν θα οδηγούσε σε δυσανάλογη γραφειοκρατία. Και εδώ εμείς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη γραφειοκρατία, όχι να δημιουργήσουμε ακόμη παραπάνω. Πρέπει ο καθένας να καταχωρεί τις ώρες εργασίας του. Δεν υπάρχει κανένας που να τον εμποδίσει γι' αυτό. Η ψηφιακή ταχογράφη δεν μπορούν να καταγράψουν τις ώρες αυτές. Ο υπάλληλο μπορεί να δείξει τις ώρες εργασία του στους, ε, στον, ε, στο αφεντικό του. Ο ε, αυτοαπασχολούμενος δεν, έχει, δεν μπορεί να δείξει τις ώρες εργασίας του σε κάποιον. Να σας θυμίσω τι γινόταν και πριν τους ταχογράφους. Όλοι οι, εργα... όλοι οι ε, οδηγοί έπρεπε να έχουν μητρό των ωρών εργασίας τους. Και αυτό βεβαίως δεν ήταν ε, μητρό τελικά, ήταν ε, τετράδιο καταγραφής πλασματικών ωρών εργασίας. Ο ταχογράφος τώρα καταγράφει τις ώρες εργασίας, το κρατήσει κάποιο το όριο των ωρών ανάπαυση που του αποδίδεται, εξαρτάται από τον ίδιο. Οι αυτοαπασχολούμενοι δεν μπορούν να ε, οδηγούν πάνω από 90 ώρε κάθε δύο εβδομάδε και πρέπει να έχουν και επαρκή χρόνο ανάπαυση. Αυτό μπορεί να γίνει και σε διασυνοριακό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε, για να μπορέσουμε να έχουμε έτσι ένα ε, ε, θεμητό ανταγωνισμό πρέπει να εφαρμοστεί σωστά σε όλη την Ευρώπη ο κανονισμός για τις ώρες οδήγηση και τις ώρες ανάπαυσης. Ο, ο αριθμός των ελέγχων θα διπλασιαστεί μέχρι το 2012 και αυτό θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να, να εξασφαλίσουμε την οδική ασφάλεια. Τώρα, ο στόχο της οδηγία είναι να, να, προστα, να προστατεύσει του εργαζόμενου. Ω εργαζόμενους. αυτό συμφωνούμε η δομή αυτή τη γραμμή ακολουθεί. Η οδηγία δίνει τη δυνατότητα να αποκλίνει κανείς από τους, από τους συνηθισμένους κανόνες μέσω των, των συλλογικών συμβάσεων και των διαπραγματεύσεων. Οπότε, ποιο θα συμφωνήσει με τις παρεκκλήσεις. Αν συμφωνήσει, δεν συνάδει με τους, με τους κανόνες. Υπάρχει ο κανονισμό για τι ώρε οδήγηση και τι ώρε ανάπαυση. Η οδηγία είναι επιπλέον νομοθετικό κείμενο για να καλύψει άλλε δραστηριότητε πέραν τη οδήγηση, α πούμε την ε, ε, φορτοεκφόρτωση κτλ. Τώρα για τον αυτοπασχολούμενο οδηγό. Ο αυτοπασχολούμενο οδηγό είναι ένα επιχειρηματία από μόνο του. Πρέπει να έχει μια, μια άδεια για να, για να λειτουργήσει η επιχείρησή του. Οπότε πρέπει να, έχει, να είναι φερέγγιο, πρέπει να ε, κάνει ελέγχου. Έτσι ώστε οι προποθέσει όλε αυτέ να πληρούνται. Και να πω επίση ότι η φερεγγιότητα είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό μπορεί να ξέρει ο αυτοαπασχολούμενος αν έχει αρκετό εισόδημα για να χρηματοδοτήσει ούτως ή την, ε, την ε, επιχείρησή του. Πρέπει να διτηρήσει και την καλή του φήμη για να, έχει την, ε, για να λάβει την άδεια του μεταφορέα. Οπότε μπαίνει στο ζύγι και η άδεια που θα έχει ένας αυτοπασχολούμενος οδηγός. Μα ενδιαφέρει η υγεία και η ασφάλεια του αυτοαπασχολούμενου. Φυσικά τον καταρτίζουμε, κάνουμε εκστρατείε μέσω οργανισμών, μέσω κυβερνητικών πρωτοβουλειών. Ε, τονίζουμε την ότι πρέπει να τρώει σωστά, να ξεκουράζεται τι ώρε που πρέπει. Όλα αυτά είναι φυσικά σημαντικά. Τώρα, το θέμα των ιονί αυτοαπασχολούμενων είναι σημαντικό και δεν είναι εύκολο να, ε, να κάνουμε το διαχωρισμό μεταξύ ενό πλασματικού αυτοαπασχολούμενου και ενό κανονικού πραγματικού αυτοαπασχολούμενου. Επίσης το θέμα το φορολογικό στις κάτω χώρες το θέμα αυτό των πλασματικών αυτοπασχολούμενων δεν είναι πρόβλημα πλέον. Γιατί υπάρχουν ε, ε, εταιρείε οι οποίε δίνουν υπεργολαβία σε μεταφορεί, οι οποίοι όμω είναι πραγματικοί αυτοποσχολούμενοι γιατί αλλιώ πρέπει η εταιρεία να καταβάλει την κοινωνική συνεισφορά για τον πλασματικό αυτοποσχολούμενο. Οπότε δεν τη συμφέρει. Φροντίζει λοιπόν να είναι όντω αυτοποσχολούμενο αυτό ο οποίο αναλαμβάνει την υπεργολαβία. Δημιουργείται λοιπόν έτσι ένας θεμητός ανταγωνισμός και αποτρέπεται η απάτη. Υπάρχει βέβαια έλλειψη οδηγών και η κατάσταση θα χειροτερέψει ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Στις ε, κάτω χώρες έχουμε και θέμα γύρενσης του πληθυσμού. Θα χρειαστούμε 8.000 νέους οδηγού κάθε χρόνο. Το ίδιο ισχύει και για τις ε, Σκανδιναβικέ χώρες, το Βέλγιο, τη Γαλλία, ακόμη και την Πολωνία. Οπότε αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείε θα προσπαθήσουν ε, να προσελκύσουν τους οδηγούς για να εργαστούν για αυτούς. Αλλά οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν και τον εργοδότη ο οποίος τους δίνει τις καλύτερες προποθέσεις εργασίας. Τώρα για την οδική ασφάλεια. Η οδική ασφάλεια συχνά χρησιμοποιείται ως λόγος γιατί θα πρέπει να καλύπτονται οι αυτοπασχολούμενοι από ε, την οδηγία. Ε, μπορείτε να ολοκληρώσετε, λέει η Πρόεδρος. Ναι, θα ήθελα να... Ε, μιλήσω για την οδηγία ασφάλεια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο πρέπει να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι οι αυτοαποσχολούμενοι είναι λιγότερο ασφαλείς από τους υπαλλήλους. Στις κάτω χώρες δημιουργήσαμε, ε, κάναμε μάλλον μια έρευνα και είδαμε ότι διακόπτει τον ομιλητή η πρόεδρος. Θα μας μιλούσατε για επιμελητή, αλλά μας μιλήσετε για άλλα πράγματα. Ο κύριος Ανδρέα, η κυρία Ανδρέα Κότσι, Κότσης έχει το λόγο, υπεύθυνη ε, της, των υποδομών στις ταχυδομικές υπηρεσίες. Έχετε το λόγο. 10 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σα πω τη δική μου άποψη. Είμαι εκπρόσωπο ε, του Συνδικάτου Βέρντι. 2,2 εκατομμύρια μέλη έχει το Συνδικάτο μας στη Γερμανία. Πριν από 7 χρόνια, οι Ευρωπαίοι νομοθέτες ήταν της άποψης ότι η ελάχιστη προϋπόθεση σε σχέση με, το, τον χρόνο εργασίας είναι απαραίτητη έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια των επαγγελματιών οδηγών. Η ασφάλεια για όλους τους εμπλεκόμενους στον χώρο αυτό θα έπρεπε να ε, αυξηθεί και να είναι πιο θεμητός ο ανταγωνισμός. Με την οδηγία 2012-2015 εφαρμόστηκαν όλα αυτά και η οδηγία αυτή ισχύει για όλους τους επαγγελματίες οδηγούς, αλλά δεν εφαρμόζεται παντού. Σε αυτά τα 7 χρόνια η κατάσταση στους ευρωπαϊκούς ε, δρόμους ε, έχει ε, αυξηθεί κατά πολύ. Ο, η, η, στρέβλος του ανταγωνισμού επίσης έχει αυξηθεί κατά πολύ. Ε, για να μπορέσουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε ε, την υγεία και την ασφάλεια ε, των οδηγών, οι οποίοι πολλές φορές είναι πάρα πολύ κουρασμένοι και πραγματικά διακυβεύεται η ασφάλειά τους και των υπολείπων οδηγών. Δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε καθόλου όλες, αυτούς τις, όλες αυτές τις προϋποθέσεις, αλλά η οδηγία αγνοεί το γεγονός ότι πέρα από, τους, από τις ώρες οδήγησης, ο οδηγός αυτός έχει και άλλη ζωή ε, πρέπει να κάνει και άλλα. Πρέπει να καθαρίσει το, το φορτηγό του, πρέπει να περιμένει, πρέπει να φορτώσει, να εκφορτώσει. Όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη. Θα ήθελα να, θέσω, να απαντήσω και στο ερώτημα για το ποιε είναι οι επιπτώσει όταν ένα ε, αυτοαπασχολούμενο ε, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Ή ποιοι είναι οι λόγοι που μόνο η τήρηση του κανονισμού 561 του 2006 ισχύει για, δεν ισχύει μάλλον για τους αυτοπασχολούμενους. Καταρχήν, μιλούμε για τον ανταγωνισμό. Προς το παρόν έχουμε μία, ένα ωράριο 48 ωρών της, ε, την εβδομάδα και ανώτατο όριο εργασίας 60 ώρες την εβδομάδα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι ώρες εργασίας για τον αυτοαπασχολούμενο μπορεί να φτάσουν τις 86. Ε, για, ε, για φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους δεν υπάρχει καμία, κανένας περιορισμός για τους ώρες οδήγησης και, και κανένα κατώτατο όριο οδήγησης. Οπότε υπάρχει απεριόριστος ο χρόνος εργασίας για τους ανθρώπους αυτούς. Οι επιπτώσεις ε, αποκλεισμού των αυτοαπασχολούμενων από το πεδίο εφαρμογής της οδηγία θα ήταν να δημιουργηθούν μικρές, ε, να, όλες αυτές οι μικρές μάλλον εταιρείες να εξαγοραστούν από μεγάλες. Η πίεση για το ελάχιστο κόστος και για, συνεχής, για συνεχή υπεροχή υπηρεσιών αυξάνεται συνεχώς. Επιπλέον, οι διάφορες οδηγίες που ε, διάφορες διαφορε... Οι διαφορές που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά και την ε, φορολόγηση και την μισθοδοσία οδηγούν σε στρέβλος του ανταγωνισμού και αυτό αυξάνεται συνεχώς. Επηρεάζονται οι ώρες εργασίας και υπάρχει φυσικά μεγάλο μειονέκτημα και για τους εργοδότες και για τους εργαζόμενους οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την ε, υπόθεση. Για τη Γερμανία τώρα. Στη Γερμανία έχουμε περίπου 54.000 ε, ε, εταιρείε που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά αγαθών. Περίπου 75%, 57% ε, απασχολείται από από, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μόνο 4% έχει πάνω από 50 εργαζόμενους. Οπότε οι περισσότεροι είναι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί οι οποίοι αποτελούν από μόνοι τους μια επιχείρηση. Η στρατηγική λοιπόν των μεγάλων επιχειρήσεων είναι να έχουμε όσο περισσότερου γίνεται αυτοπασχολούμενου οδηγού. Μερικά παραδείγματα γι' αυτό. Σένκα, μια μεγάλη εταιρεία που έχει έδρα στην ε, Γερμανία, στι αρχέ του χρόνου έκανε τους υπαλλήλους της αυτοπασχολούμενους με, το ίδιο, ε, με τις ίδιες συνθήκες και με την, ίδια, ε, με την προσφορά να χρονομισθώνει κανείς το, το φορτηγό. Επίσης, άλλη μεγάλη εταιρεία που έχει έδρα σε τέσσερι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Ε, η ε, Αγκουστίν που έχει έδρα στην Αυστρία. Επίσης, μετέτρεψε τους ε, υπαλλήλου τη σε αυτοαπασχολούμενου. Όλη αυτή η κατάσταση πραγματικά οξύνει την κατάσταση και δεδομένη και τη οικονομική κρίση. 25 με 30% μείωση του κύκλου εργασιών, αφαιρεγγιότητα των, μεγάλων, των μικρών επιχειρήσεων. Συγγνώμη. Αυτό οδηγεί στο ότι μόνο και μόνο για το θέμα του κόστους υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον ανταγωνισμό. Πάω τώρα στις συνθήκες εργασίας και στην ε, ασφάλεια και την υγεία των ε, οδηγών. Το, ο κίνδυνος ε, ο κίνδυνο ατυχημάτων αυξάνεται από την 8η ώρα οδήγηση και πραγματικά αυξάνεται πάρα πολύ μετά την 9η ώρα. Αν κάποιο είναι 10 ώρε ξύπνιο, η απόδοσή του μειώνεται δραστικά. Το όριο σε περίπτωση ε, αλκοτέστ είναι 0,5 στις περισσότερες, στις περισσότερες χώρες, αλλά ε, σε πάρα πολλές οι οδηγοί ξεπερνούν το 1 ε, χιλιογραμμάριο. Οι επιπτώσεις λοιπόν όλων αυτών των μεγάλων, των μακρών ωρών εργασίας ε, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ακόμη και ένα δευτερόλεπτο να, να τον πάρει ο ύπνος τον οδηγό πραγματικά μπορεί να οδηγήσει σε, θανάσιμες, ε, σε θανάσιμα προβλήματα, σε ατυχήματα, σε, στη, ε, αμφισβήτηση και τη δική του ασφάλειας και των υπολείπων οδηγών που βρίσκονται στον δρόμο. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη μεγάλη για ελέγχου βεβαίως Αυτό φέρνει μαζί του και μεγάλο άχθος. Πολλέ φορέ ε, στου ελέγχου αυτού εμπλέκονται και πάρα πολλέ ε, αρχέ. Δηλαδή, η οικονομική αρχή που είναι υπεύθυνη για την, ε, για την οντότητα, την επιχείρηση αυτή καθ' αυτή. Η, το Υπουργείο Εργασία για τι ώρε εργασία του, του οδηγού. Όλες Όλε αυτέ οι διαφορετικέ όμω αρχέ εμπλέκουν μπλέκουν περισσότερο τα πράγματα από ότι τα διευκολύνουν. Είναι λοιπόν πραγματικά πολύ σοβαρή η κατάσταση. Ε, το Υπουργείο διαπιστώνει ότι οι παραβιάσει έναντι αυτών των κοινωνικών προϋποθέσεων αποτελούν ένα πολύ μεγάλο παράγοντα πρόκλησης ατυχημάτων. Υπάρχει λοιπόν μεγάλος συσχετισμός μεταξύ των ατυχημάτων, του κινδύνου πρόκλησης ατυχημάτων και των όρων εργασίας. Το 2001 έγινε μία έρευνα την οποία θέλω να σας θυμίσω για την κούραση. Η κούραση αποτελεί τον παράγοντα για 20% των ατυχημάτων. Αλλά η κούραση δεν θεωρείται, ε, ε, η κούραση μάλλον δεν αποτελεί παράγοντα ε, όταν λαμβάνεται υπόψη το ωράριο εργασίας. 50% των ερωτηθέντων οδηγών ε, πραγματικά είπαν ότι μπορεί να τους πάρει ο ύπνος για δύο δευτερόλεπτα, για τρία δευτερόλεπτα. Αυτό ξάνεται τον, ε, τη νύχτα και όταν ε, είναι άτακτο το ωράριό τους. Η ασφάλεια, όπως λέει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Οδική Ασφάλεια, συνήθω μπαίνει στην άκρη όταν υπάρχει η εμπορική λογική. Ότι η μεταφορά ας πούμε, των ατόμων και των αγαθών πρέπει να είναι ευέλικτη, πρέπει να γίνεται 24 ώρες το 24ωρο, δεν πρέπει να υπάρχουν ε, ε, προσκόμματα αλλά η εργασία έχει να κάνει, οι ώρες εργασίας έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια του ε, οδηγού. Στην ε, Ευρώπη πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ των οικονομικών ε, παραγόντων και των κοινωνικών προϋποθέσεων. Δεν μπορούμε να, πηγαίνει, να είναι, δεν μπορεί να γέρνει μονόπαντα η ζυγαριά. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει θεμητό ανταγωνισμός, σωστέ προποθέσει προϋποθέσεις για την μεταφορά αγαθών και προσώπων, καλύτερες συνθήκε εργασία, καλύτερη προστασία για όλους τους επαγγελματίες οδηγού και καλύτερη ασφάλεια για όλους όσους εμπλέκονται στον τομέα αυτό στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν και οι ώρες, και η οδηγία που αφορά τις ώρες εργασία πρέπει να, εφαρμοστεί, πρέπει να υπάρξουν οι ίδιες συνθήκες. Ο διαχωρισμό τώρα μεταξύ των ιονί και των κανονικών αυτοαπασχολούμενων ε, μπορεί να γίνει μόνο σε μεμονωμένε περιπτώσει. Οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να εφαρμόζουν, μάλλον πρέπει για τους αυτοαπασχολούμενους να εφαρμόζεται η οδηγία για, τα, ε, για, την, ε, για το ωράριο εργασίας Αυτό θα αποτελούσε μεγάλη συμβολή στο να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, όλοι είχατε γραπτά την παρουσίασή σας, λοιπόν παρακαλώ να τη δώσετε στη γραμματεία ώστε να μπορέσουμε να τα διανύμουν στα μέλη και σε αυτούς που δεν ήταν παρόντες. Έχουμε 10 λεπτά και τέρμα. Έχω πέντε που θέλουν τον λόγο. Ενάμιση λεπτό ο καθένας. Εκτός αν υπάρχει κι άλλο που θέλει να παρέμβει. Ένα λεπτό ο καθένας λοιπόν. Στην αρχή η συγκητρία ή στο τέλος θέλει το λόγο. Αρχή ή τέλος κυρία Μπάουερ. At the end. Okay, στο τέλος. Σαν συμπέρασμα ή έχετε ερωτήσει, κυρία Μπάουερ. Στο τέλος. Ωραία. Χαιρετίζω και τους επισκέπτες της κυρίας Κώστα. Δεν μπορέσαμε να απευθυνθούμε σε αυτούς, αλλά φύγανε εντωμεταξύ οι περισσότεροι. Ένα λεπτό ο κάθε μιλητής. Κυρία Ευλίν Ρενιέ, ο κύριος Βαντάλεν. Ε, θα τελειώσουμε αγγλογαλλικά υποχρεωτικά. Ο κύριος Βαντάλεν. Κυρία Ρενιέ πρώτα. Λυπούμε καταρχήν που προφανώς κανένας δεν είναι εδώ από τους ε, Ευρωπαίους, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εργαζομένων. Εργοδοτών, συγγνώμη. Ε, εργοδότες δηλαδή που παίρνουν μέρος στον κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την καλύτερη διακυβέρνηση τώρα. Euh, impressionné. Poursuivez votre propos. Vous ah Ένα λεπτό έχετε, κύριε Λοιπόν, είπατε για τους ε, ψηφιακούς, ε, ε, για, το, για τους ψηφιακούς χάρτες. Να σας θυμίσω την έκθεση Στόιμπερ. Εκεί είχε ζητηθεί να γίνουν εξαιρέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτή τη συζήτηση νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να συμπεριληφθεί. Γιατί αναφέρθηκε η σωστή μέτρηση οδήγησης και ανάπαυσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους αυτοπασχολούμενους και για τους ιονή αυτοπασχολούμενους, αλλά και για τους κανονικούς αυτο, ε, υπαλλήλους να συμπεριλαμβάνονται οι ε, οδηγοί. Ο κύριος Πίτερ Βαντάλεν και μετά η κυρία Μάρτιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο συγκεκριμένα σημεία θα ήθελα να στήξω. Θα ήθελα να ζητήσω από τους ομιλητές να επανέλθουν σε αυτό που είπε ο κύριος Κράμερ στην αρχή της παρέμβασής τους. Γιατί οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να εντάσσονται σε αυτή την οδηγία αφού ποτέ δεν είχε συμβεί αυτό κατά το παρελθόν. Μπορεί κάποιο να απαντήσει σα παρακαλώ σε αυτή την ερώτηση του κυρίου Κράμερ. Δεύτερο σχόλιο. Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλέ ενώσει αυτοαπασχολούμενων στις εσωτερικές πλωτές ε, μεταφορές παραδείγματος χάρη. Χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι που τηρούν την, ε, τις ρυθμίσεις για τον χρόνο εργασίας. Διότι ένα ατύχημα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σημαίνει γιόκα εργασία, πολλές ζημιές, πολλές δεπάνες. Συνεπώς είναι ένας παραλληλισμός που μπορούμε να σεβαστούμε και να ακολουθήσουμε. Η κυρία Μάρτιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ασφάλεια. Τα στοιχεία δεν υποστηρίζουν την... το γεγονός ότι θεωρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι μεγαλύτερος κίνδυνος. Κανένας δεν μας έχει δώσει τέτοιες πληροφορίες. Και η νομοθεσία που περνάει από το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να βασίζεται σε σωστά στοιχεία, όχι σε υποθέσεις. Αν πάρουμε την οδική ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας, στον οδικό τομέα λιγότερο από 5% εμφάνισαν πρόβλημα. Λοιπόν, δεν είναι όλες οι στατιστικές καλές, κακές, με συγχωρείτε. Ας χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία. Οι αυτοαπασχολούμενοι είναι ένα θέμα, αλλά δεν πρέπει, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Εδώ θα λύσουμε ένα πρόβλημα και θα δημιουργήσουμε ένα άλλο η λύση για τους αυτοαπασχολούμενους δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να ενταχθούν σε αυτή την οδηγία. Η γράφει τώρα. Πώς μπορούμε ε, να μετρήσουμε το χρόνο των αυτοαπασχολούμενων. Ε, ε, έχουμε επιθεωρητές να παρακολουθήσουν τον κάθε οδηγό όταν πηγαίνει σπιτάκι του, όταν έρχεται σε επαφή με οτιδήποτε κτλ. Η κυρία Μωρά. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που οργανώσατε αυτές τις ακροάσεις. Μας φωτίζουν πρέπει να σας πω και μας οδηγούν να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας. Είμαστε στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Υπήρξαν πολλές μαρτυρίες, διαφορετικές απόψεις και δουλειά μας είναι να προχωρήσει η κοινωνική Ευρώπη. Δεν μπορούμε να δεχθούμε να υπάρξουν αποφάσεις οι οποίες θα είναι αντίθετες από, με μια οδηγία που ισχύει από 23 Μαρτίου και δεν μπορούμε να δεχθούμε οπισθοδρομήσεις. Κυρία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Φαίνεται ότι πραγματικά οι τοποθετήσει μας βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση. Αλλά το θέμα που έθεσε η συνάδελφος ακριβώς είναι το βασικό. Ε, το να έχουμε μια οδηγία η οποία δεν τηρείται δεν οδηγεί πουθενά. Στην οδηγία προβλέπεται ότι αυτό απασχολούμενοι ε, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή της οδηγίας. Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά δεν είναι εφικτά. Λοιπόν, το πρόβλημα προκύπτει από τη μη πρακτικότητα του μέτρου. Πιστεύω λοιπόν ότι οι εμπειρίες που αναφέρθηκαν εδώ ε, είναι σαφέστατες. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Τούρινεν και Χάντελ, αλλά έχουν ήδη λάβει το λόγο. Δεν θα τους δώσω το λόγο. Ε, τώρα, η κυρία Γιώργενσεν. Κυρία Πρόεδρε, Μία ερώτηση. Με τον τρόπο αυτό, με συγχωρείτε, υπήρξε ένα πρόβλημα τεχνικό μεταξύ καμπινών και χάθηκε η διερμηνία κάπου στο δρόμο η πρόεδρος και η γαλλική διερμηνία ε, έχασε λίγο τα νερά της. Πολύ ίντομα λοιπόν. Ε, με σωστά γαλλικά αυτή τη φορά. Να μπορούμε να διαλέξουμε δύο σωστά πράγματα. Ε, ή ένα καλό και ένα άσχημο. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται ε, σε σχέση με την οδική ασφάλεια είναι το εξής. Μπορούμε να διαλέξουμε να έχουμε ένα καλύτερο έλεγχο του χρόνου ανάπαυσης. Ή ε, προτιμάμε να έχουμε αυτοαπασχολούμενους μόνιμα. Ευχαριστώ. Ζητώ από τους δύο προσκεκλημένους να τηρήσουν τους ίδιους κανόνες. Δύο λεπτά. Τον τελευταίο λόγο θα τον έχει η εισηγήτρια. Κύριε Κότσιτς. Το ερώτημα που τέθη ήταν γιατί ξαφνικά εμπίπτουν σε αυτήν ή θα έπρεπε να εμπίπτουν σε αυτήν την οδηγία ή α, αυτοαπασχολούμενοι. Το θέμα αυτό έχει που το συζητούμε εδώ και χρόνια. Η οδηγία εφαρμόστηκε και τώρα πρέπει να ε, ε, υποβλήθηκε και πρέπει να εφαρμοστεί οι αυτοαπασχολούμενοι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με τους υπαλλήλου. Δεν είναι καινούριο αυτό. Ήδη το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Οπότε πρέπει να πω ότι οι αυτοαπασχολούμενοι στις οδικές μεταφορές δεν, είναι, δεν αποτελούν μεγαλύτερο κίνδυνο από τους υπαλλήλους, αλλά όταν, όταν δουλεύουν τόσο πολλές ώρες αποτελούν και αυτοί κίνδυνο. Δεν μιλούμε για λιγότερο κίνδυνο ή περισσότερο κίνδυνο. Δεν προσπαθούμε να ζυγίσουμε τον κίνδυνο. Προσπαθούμε να πούμε ότι αυτοί οι επαγγελματίε οδηγοί, είτε είναι, είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι, είτε είναι ε, υπάλληλοι, πρέπει να, να έχουν ένα συγκεκριμένο ωράριο. Πρέπει να περιορίζονται οι ώρε εργασία του. Γιατί αλλιώ αποτελούν κίνδυνο. αντιμετωπίζουν δηλαδή τον ίδιο, ε, το, αποτελούν το ίδιο πρόβλημα και με έναν απλό οδηγό που είναι πολλές ώρες στο τιμόνι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κράμερ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, γιατί να υπαχθούν στην οδηγία οι ανεξάρτητοι. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Και θα σας το πω πριν με κόψετε. Τα τελευταία χρόνια, από το 97 και μετά, υπάρχει μόνο καλύτερη ασφάλεια οδικών, οδική, οδική ασφάλεια και υπάρχει τεκμηρίωση για τη βελτίωση της κατάστασης. Επίσης, η, το, το εμπόρευμα είναι ασφαλέστερο και άρα έχουμε χαμηλότερο αριθμό ατυχημάτων και χαμηλότερο αριθμό θυμάτων. Τώρα, για την επιλογή, ανεξάρτητη εργαζόμενη ή αυστηρότερη έλεγχη. Εγώ θα επέλεγα για τις δύο δυνατότητες όχι μόνο τη βελτίωση των ελέγχων για το, χώρο, για το χρόνο εργασίας. Θα επέλεγα, θα κάλυπτα και τους μισθωτούς εργαζόμενους οδηγούς. Και αυτό βελτιώνει την κατάσταση. Όταν ε, η οδηγία εφαρμόζεται, το ερώτημα που τίθεται είναι μπορούμε, όχι αν καλύπτουμε τους ανεξάρτητους ή όχι, αλλά κατά πόσον πρέπει να τους καλύψουμε ή όχι. Έχει την Επιτροπή και λέει θα κάνουμε μία πρόταση και η οδηγία θα μπορεί να προχωρήσει ε, εκτενέστερα. Αυτό δεν είναι σωστό. Ευχαριστώ η κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Δεν ξέρω να... ίσως να έχω χρόνο για μια σύντομη περίληψη. Πήραμε πολλά στοιχεία, όχι κατά ανάγκη συναφή με την οδηγία. Η οδηγία αφορά οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Όπως και η 561. Να σας πω την αλήθεια, με απογοήτευσε το ότι ε, ακούγονται πολλά στοιχεία και νούμερα. Η οδηγία του 2002 μεγιστοποιεί σε τέσσερις μήνες την προθεσμία.